Ja, Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά. Και πάμε στο επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη που είναι ανταλλαγή απόψε με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γύρκη Κατάινεν. Ως αντιπρόεδρος είναι αρμόδιος για την απασχόληση και την ανάπτυξη, άρα και τα μεγάλα θέματα ανταγωνισμού για τις μεταφορές, επενδύσεων και τα λοιπά και ανταγωνιστικότητας. Και βεβαίως για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εκεί ε, ε, βρίσκεται πλέον και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, το λεγόμενο ΕΦΣΥ, και τις επόμενες μέρες θα συζητήσουμε για παράταση της διαρκείας του Ταμείου αυτού. Ο κύριος Κατάινεν θα μας ε, παρουσιάσει σήμερα τους στόχους ε, και τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές και τον τουρισμό και ε, για σήμερα και για το μέλλον. Χαίρομαι που είστε παρόν, χαίρομαι που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Καλωσορίσατε θερμά όπως πάντα. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την δυνατότητα να συζητήσουμε τα θέματα αυτά μαζί σας. Είχα σκοπό να συζητήσουμε περισσότερο για το ΕΦΖΙ, ΕΦΣΙ με συγχωρείτε 1,0 και, και 2,0, όπως επίσης και ε, για τα παραπλευρά στοιχεία του επενδυτικού ε, αυτού πακέτου, αλλά ίσως είναι καλύτερο να ξεκινήσω με κάποια αριθμητικά δεδομένα, γιατί πριν από 1,5 χρόνο κάναμε μια συζήτηση με την Επιτροπή σας όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την ε, πρόταση ε, για την χρήση αυτών των κονδυλίων για την κεφαλαιοποίηση του ΕΦΣΙ και ξέρω ότι ίσως δεν ήσασταν πάρα πολύ θερμοί. Λοιπόν, από τότε που ξεκίνησε το ΕΦΣΙ, να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Για τα έργα στον τομέα των μεταφορών έχουμε χρηματοδοτήσει επενδύσεις που τελικά με τη μόχλευση έφτασαν τα 11 δις. Άρα λοιπόν σε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο για, το, για τις μεταφορές το πλεονέκτημα ήταν 11 δις. Κοιτάξαμε και σε πόσα δάνεια ή χρηματοδότηση έχουν χορηγηθεί από το ΕΦΣΙ στις μεταφορές έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε τα 11 ε, δις αυτά της α, ε, ε, μόχλευσης. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε με 2 δις τα οποία μόχλευσαν 11. 11 δις σε επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών. Δηλαδή, είναι όλο το ποσό που πήραμε από το μηχανισμό. Άρα λοιπόν η πρόταση που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσθέσουμε 1,1 δις σε αυτές τις πιστώσεις του μηχανισμού και αυτό το 1,1 δις να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε μαζί με το ΕΦΣΙ να χρησιμοποιηθεί για να επενδύσουμε σε ε, έργα υποδομής. Εάν λοιπόν υπολογίσουμε τις απώλειες αυτό το οποίο θα καταλήξουμε είναι πως τελικά ε, κερδίσατε πολύ περισσότερα από ό,τι χάσατε από το, από το μηχανισμό Connecting Europe και τελικά είσαστε καλύτερη θέση από ό,τι ήσασταν πριν ξεκινήσει το ΕΦΣΙ. Έχετε χρηματοδοτήσει μέσω των εργαλείων όλες αυτές τις επενδύσεις και αυτό το οποίο αποκομίσαμε και από τους ενδιαφερόμενους και από την αγορά είναι ε, πως τα δάνεια τα δάνεια του Connecting Europe είναι λιγότερο ελκυστικά από αυτά που γίνονται στα πλαίσια του ΕΦΣΥ. Άρα λοιπόν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΦΣΥ είναι και αυτά πιο ελκυστικά από τα ε, χρηματοδοτικά εργαλεία του μηχανισμού Connecting Europe. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί το ΕΦΣΥ μπορεί να ε, μοχλεύσει τελικά τα ίδια ποσά, αλλά με πιο θετικές ε, ροές. Όπως γνωρίζουμε, Είμαστε στον τέταρτο χρόνο της ανάκαμψης της οικονομίας μας, αλλά ακόμα οι ρυθμοί είναι εξαιρετικά ε, χαμηλοί και επίσης για την ανάπτυξη οι μεσομακροπρόθεσμες προβλέψεις είναι αρκετά χαμηλές, άρα λοιπόν οι επενδύσεις δεν είναι αρκετές. Ε, το ΕΦΣΙ δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο ολόκληρο, αλλά το καλύτερο εναλλακτικό σενάριο θα μπορούσε να συνεισφέρει για να καλύψει τουλάχιστον το 1 τρίτο των απαραίτητων επενδύσεων. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θα ανακουφίσει κατά το 1 τρίτο το, την οδύνη την οποία έχουμε χρειαστεί να ε, υποστούμε και δεν έχει να κάνει αυτό τόσο πολύ με το γεγονός ότι λείπουν τα κονδύλια. Όχι, οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή έχουν καθυστερήσει γιατί υπάρχουν και διαστροτικά προβλήματα. Το ΕΦΣΥ πρέπει να σου πω ότι παραδίδει ε, τα όσα έχει υποσχεθεί και όχι μόνο σε επίπεδο αριθμών με επενδύσεις που έχουν εγκριθεί και που έχουν φτάσει τα 138 δις σε 27 κράτη-μέλη. Όχι, 27 κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν το ΕΦΣΙ για διάφορους ε, λόγους με χρηματοδότηση που έχει φτάσει στα 138 δις σε επενδύσεις, το οποίο σημαίνει ότι ε, έχουμε ε, καταφέρει να χρηματοδοτήσουμε και επενδύσεις που δεν θα είχαν χρηματοδοτηθεί χωρίς αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Πρέπει να σας πω πως έχει χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει συγκεράσει και την εμπειρία της ΕΤΕ και την εμπειρία τη δική μας με αποτέλεσμα με πιο ευφυή κατανομή των πόρων που έχουμε που δεν είναι απεριόριστοι δίνοντας ε, θετικά μηνύματα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Στα σκαριά αυτή τη στιγμή έχουμε 16 ε, ή με συγχωρείτε 60 16, 16 εγκεκριμένα project, εκ των οποίων τα 5 είναι τη στιγμή της υπογραφής. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό ε, ε δυναμικών επενδύσεων που θα φτάσει στα 11 δις. Να σας πω πως έχουμε και διάφορα ε, σχέδια τα οποία είναι στη φάση της προέγκρισης που πιθανώς θα κινητοποιήσουν επενδύσεις της τάξης του, 3, του ύψους του 3,5 δις. Για τον κλάδο των μεταφορών να σας πω πως έχουμε μία πλατφόρμα ΕΦΗ e που θα επιταχύνει τις επενδύσεις έτσι ώστε να ε, έχουμε λιμάνια στην Ισπανία, τρένα στην Ιταλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο και εγκαταστάσεις σχετικές με αυτά τα δίκτυα και ένα πολύ μεγάλο project στη Σλοβακία, όπως επίσης και αρκετές υποδομές, έτσι ώστε να καλύψουμε, σας ε, ε, επαναλαμβάνω, επενδυτικά κενά σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε επίσης κάποια εργαλεία που έχουν ως σκοπό να φέρουν τα επενδυτικά αυτά έργα σε πέρας. Έχουμε λοιπόν ε, το hub που έχει ως σκοπό να προωθεί αυτά τα έργα και που προσφέρει 365 μέρες το χρόνο τεχνική βοήθεια έτσι ώστε σε όποια χώρα και να έχει κανείς ένα project να μπορεί να το στήσει και να ξεκινήσει. Και μέσω των ε, τεχνικών συμβουλών μπορεί κανείς να βρει και ποιες είναι οι κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης. Αυτό το hub, αυτός ο ο κόμβο έχει αντιμετωπίσει 257 αιτήματα βοήθεια από όλα τα κράτη-μέλη και πρέπει να σα πω πω στο website, ε, στην διαδικτυακή πύλη αυτού του hub υπάρχουν πάρα πολλέ πληροφορίε και θα σα παρατρύνω να ανατρέξετε σε αυτέ, γιατί πάρα πολλέ πληροφορίε θα αντλήσετε που ενδεχομένω θα σα είναι χρήσιμε και πιστεύω ότι θα πρέπει και η εκλογική σα ε, περιφέρεια να ενημερωθεί για αυτή τη δυνατότητα τεχνική βοήθεια που δίνεται μέσω του hub, του Advisory Hub γιατί πολλές φορές και οι εθνικές διοικήσεις χρειάζονται συμβουλές για το πώς μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα ενός έργου και μπορούν να το κάνουν μέσω του website της ιστοσελίδας δηλαδή του Hub. Επίσης πρέπει να σας πω πως είναι πολλά υποσχόμενο το γεγονός πω πάρα πολλά από αυτά τα αιτήματα που καταφθάνουν είναι αιτήματα του ιδιωτικού κλάδου, ο οποίο προφανώς έχει δείξει πως για να ενισχυθεί η ποιότητα των έργων χρειάζονται ενημέρωση, ενημέρωση που θα δοθεί από τι δικέ μας υπηρεσίες. Ένα ακόμα θέμα ε, για το οποίο θα ήθελα να σας παροτρύνω να κάνετε προσπάθειες είναι το πόρταλ που έχουμε, διαδικτυακή πύλη ε, για τα ευρωπαϊκά έργα. Και να σας πω πως εκεί έχουμε 121 έργα από διάφορα κράτη-μέλη και αυτή η διαδικτυακή πύλη, αυτό το πόρταλ είναι σαν ένα σύστημα ραντεβού online ε, dating online δηλαδή. Φέρνει σε επαφή τους επενδυτές με τα κονδύλια. Και ξέρετε πως τα πιο, ε, οι πιο πολλές επισκέψεις έχουν γίνει για ελληνικά project σε αυτή την ε, πύλη. Και τέσσερα στα πέντε είναι ε, υποδομές. Οπότε ε, προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Ελλάδα για τις υποδομές. Και θα ήθελα να ρίξετε κι εσείς μια, μακριά, μια ματιά. Εγώ πήγα και στο Χονγκ Κονγκ και στην Νότιο Κορέα και στην Ιαπωνία και στη Σιγκαπούρη και όποτε πηγαίνω στα μέρη αυτά προσπαθώ να έρθω σε επαφή με επενδυτές και κυρίως με όσους επενδύουν σε υποδομές. Και για μένα ήταν αρκετά ενδιαφέρον να αναγνωρίσω και να ακούσω αυτό που μου λένε. Δηλαδή ότι ήδη βρήκαν βρήκαν το πόρταλ αυτό, τη διαδικτυακή πύλη για τα ευρωπαϊκά project και πολλέ φορέ λένε ότι είναι οι πρώτοι που μπαίνουν γιατί θέλουν να βρουν το πιο ενδιαφέρον project πρώτοι. Και κάποια από αυτά, για παράδειγμα, κάποιοι από αυτού στο Hong Kong ήδη προετοίμασαν κάποια από τα ελληνικά. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό με ικανοποίησε ιδιαίτερως. Λοιπόν, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή αυτή πύλη και θα σας δώσει μια πολύ ε, πλήρη εντύπωση για το πώς λειτουργεί και στείλτε το μήνυμα αυτό στην εκλογική σας περιφέρεια. Υπάρχουν δήμοι, υπάρχουν ε, κυβερνητικές αρχές που να θέλουν να επενδύσουν. Μήπως είναι ιδιωτικό κλάδος που χρειάζεται να επενδύσει. Και να στείλει στη διαδικτυακή μας πύλη αυτό το έργο έτσι ώστε να είναι πιο ορατό και να σας πω πως θέλουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ επενδυτών και να σας πω πως είναι πολύ χρήσιμο το εργαλείο αλλά δεν χρησιμοποιείται επαρκώς. Χρειαζόμαστε λοιπόν και γι' αυτό σας παροτρύνουμε να επισκεφτείτε αυτή τη διαδικτυακή πύλη, σας επαναλαμβάνω για τα πολλά και ενδιαφέροντα που θα βρείτε εκεί. Τώρα, επενδυτική Κλαδί και ε, τι γίνεται με τα εμπόδια για την επένδυση και πώς μπορούμε αυτά να τα ξεπεράσουμε. Όλοι χρειαζόμαστε ένα προβλέψιμο και σταθερό κανονιστικό περιβάλλον και ξέρουμε ότι έχουμε μια σειρά από συγκεκριμένα ε, βήματα τα οποία έχουμε πάρει σε λιγότερο από δύο χρόνια που είναι πολύ σημαντικά για τον κλάδο των μεταφορών. Η Eurostat, όπως επίσης και το ε, κέντρο πραγματογνωμοσύνης της ΕΤΕ που στις 29 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε μια κατευθυντήρια γραμμή που ξεκι... καθαρίζει κάποια θέματα για την τήρηση των εθνικών λογαριασμών και για το πώς ε, θα πρέπει να καταχωρούνται τα ΣΔΙΤ έτσι ώστε να ξέρουμε αν πρόκειται για στοιχεία εντός ή εκτός ισολογισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα κράτη-μέλη και πρέπει να σας πω πως έχουμε μειώσει ε, και τις χρεώσεις για αυτές τις επενδύσεις στην, και τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις για αυτές τις επενδύσεις σε υποδομές. Με ποιο τρόπο? μειώνοντας, μειώνοντας τα όσο χρειάζονται να κάνουν οι ασφαλιστικές στον χώρο αυτό κατά 30% εάν επενδύουν σε υποδομές. Το οποίο σημαίνει ότι έχει απελευθερωθεί γύρω στα 20 εκατομμύρια ε, 20 δις ε, σε κεφάλαια που μπορούν πια να μπουν στην αγορά. Προσπάθησαμε να ευθυγραμμίσουμε και κάποιες διαδικασίες, να τις επισπεύσουμε, δηλαδή ε, κρατικές προμήθειες, κρατικές ενισχύσεις και το κατά πόσο θα πρέπει να μειώσουμε και ε, τις χρεώσεις προς τις τράπεζες οι οποίες αναλαμβάνουν ε, ε κάποιους κινδύνους αυτές τις επενδύσεις και όπου πρέπει να δούμε αν χρειάζεται να μειώσουμε καθόλου τα επίπεδα ε, που έχουμε εντάξει ε, στους σχετικούς κανονισμούς και κυρίως στο πακέτο της Βασιλείας. Έτσι λοιπόν με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να επενδύσουν και έχουμε και συστάσεις ανακράτως για μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο χώρο των επενδύσεων. Αυτές οι, επενδύσεις, αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι ένα προαπαιτούμενο έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερα επίπεδα επενδύσεων στα κράτη-μέλη. Μετά για το ΕΦΣΙ 2,0. Λοιπόν, το ΕΦΣΙ και το σχέδιο το επενδυτικό είναι η αρχή μιας μετακίνησης στην πολιτική μας για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε για να προσελκύσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις στην χρηματοδότηση των υποδομών στην κοινοτομία και στις μικρομεσαίες στην ε, Ευρώπη. Και γι' αυτό έχουμε προτείνει να επεκταθεί το ΕΦΣΙ και σε διάρκεια και σε οικονομική ε, και σε κεφαλαιοποίηση. Πιστεύουμε πως με αυτή την επέκταση θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε, να μοχλεύσουμε τουλάχιστον ε, τρει ευρώ σε επενδύσεις μέχρι τα τέλη του 2020. Και ε, για να ενισχύσουμε το κομμάτι που είναι εγγυήσει, έχουμε ζητήσει να μας δοθεί 155, ε, ένα κεφάλαιο 155 εκατομμυρίων ευρώ από το μηχανισμό Connecting Europe, ε, έτσι ώστε να το προσθέσουμε στο φάκελο για τις επιχορηγήσεις ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Και έχουμε προτείνει, θα πρέπει να δουλεύει το ΕΦΣΙ εγκάρσια για να πετύχουμε και τους στόχους της COP21 και να επιτρέψει να γίνει η μετάβαση σε μια σε χαμηλής εκπομπές άνθρακα οικονομία με πιο εύκολο τρόπο. Ατενίζοντας το μέλλον, επίσης αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με την ΕΤΕ για να παραδώσουμε νέα οικονομικά προϊόντα, νέες λύσεις και να στοχεύσουμε τη στήριξη στις νέες, ε, στους νέους βιομηχανικούς κλάδους και στου νέου οικονομικού κλάδου με τον ίδιο τρόπο στα 28 κράτη-μέλη και βέβαια να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και τις, ε, ε, τα λάθη τη αγορά σε κάποιου ε, κλάδου των μεταφορών. Πρέπει να σα πω ότι τα οικονομικά αυτά οχήματα θα μπορούσαν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να στηρίξουν την ψηφιοποίηση, για παράδειγμα, τα καθαρότερα οχήματα που θα έχουμε στο σύστημα διαχείριση ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Όμω, πρέπει να σα πω πω είναι προβληματική η χρηματοδότηση των project για τις μεταφορές, γιατί δεν μπορούν να χρηματοδοτούν μόνο από το ΕΦΣΥ ή από κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο μόνο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συγχωνεύσουμε αυτέ τι επιχορηγήσει με κάποιο είδου επιπλέον χρηματοδότηση και ιδιωτική χρηματοδότηση και θέλουμε να γίνει μια μεταφορά 1,1 δις κονδυλίων από το Connecting Europe Facility έτσι ώστε όλα αυτά να αναμειχθούν και να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε κάποια έργα από τα TEN τα οποία έχουν υψηλή κοινωνικο-οικονομική σημασία έτσι ώστε να ξεπεράσουμε την έλλειψη στη χρηματοδότηση με τη μόχλευση που θα κάνει το ΕΦΣΙ ως καταλήτης δημιουργώντας, δημιουργώντας μια ε, βέλτιστη προσέγγιση έτσι ώστε να ε, δρέψουμε τα πλεονεκτήματα και των δύο κόσμων του ο κόσμου της ιδιωτικής χρηματοδότησης και της δημόσιας χρηματοδότησης. Αυτή λοιπόν η ανάμειξη, αυτό το blending θα πρέπει να επιταχύνει την εκτέλεση των έργων και να διευρύνει αυτά τα οποία έχουμε ήδη στα σκαριά. Και πρέπει να σας πω πως υπάρχει και το γεωγραφικό ε, στοιχείο το οποίο θα πρέπει να καλύψουμε και ε, για το hub που έχουμε, το advisory hub, θα πρέπει αυτό να κάνει παραπάνω προσπάθειες έτσι ώστε μέσω των υπηρεσιών της ΕΤΕ να καταφέρει να εξαλείψει την ισορροπία που υπάρχουν μεταξύ των κρατών συνοχής και μη συνοχής. Θα κλείσω εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι γιατί η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε με το ΕΦΣΥ είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Και ξέρετε πως υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη όπου πολλοί θα έπρεπε να γνωρίζουν το ΕΦΣΥ και δεν το γνωρίζουν. Έχω ταξιδέψει σε όλα τα κράτη-μέλη και πρέπει να σας πω πως κάθε μέρα, κάθε μέρα εγώ διαφημίζω το ΕΦΣΥ. Εγώ χρειάζομαι όμω τη βοήθειά σα. Εσεί ξέρετε Ποιε είναι οι ανάγκε σα. Και εσεί θα πρέπει να με στηρίξετε και σε κάθε εκδήλωση που οργανώνετε θα πρέπει να μιλάτε για το ΕΦΣΥ, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να ε, σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν μπούμε τώρα στη συζήτηση με ερωτήσει και απαντήσει, θα ήθελα να καλωσορίσω ε, μια ομάδα επισκεπτών από τη Βάδη Βιρτεμβέργη, το τοπικό Υπουργείο Μεταφορών. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας και στις συζητήσεις μας. Κύριος Κατάινεν θα φύγει να πάει στην Ινδία παρακαλώ και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πρώτα οι συντονιστές τρία λεπτά και μετά τα μέλη ένα λεπτό έκαστος για τις ερωτήσεις. Ο Βιμ Φαντεγκάμπ πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε πάρα πολύ. Και για το γεγονός ότι ο Επίτροπος ήρθε στην Επιτροπή Μεταφορών σε ένα ιδιαίτερο έτσι, χρονικό σημείο ε, σήμερα. Ο συνάδελφος Πίπερ θα κάνει και εκείνος κάποιες παρατηρήσεις, αλλά εγώ ο συντονιστής να πω μερικά πράγματα. Πρώτον, για τα χρήματα από το ΣΕΦ, το Connecting Europe Facility τη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη που πήγανε στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ακούγεται επιτυχία ότι 2,2 δισεκατομμύρια βάλαμε εκεί και η μόχληψη έφτασε στα 11,1 ε, στις επενδύσεις από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ωραία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μας πονάει λιγότερο, γιατί εμείς δώσαμε όλα αυτά τα λεφτά. Μαζί με τον ορίζοντα 2020, ως Επιτροπή Μεταφορών, έπρεπε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και να πάει από το ΣΕΦ στην ΕΦΣΗ. Δεν το πήρατε από τη Γεωργία ε, αυτό το κονδύλι, ούτε από τη Συνοχή, ε, αλλά από τις μεταφορές παρακαλώ. Και για μας παραμένει ένα αγκάθι αυτό και δύσκολη αφετηρία. Πολύ ωραία ε, βιβλία γράφεται για την επιτυχία του Ταμείου Στατιδικών Επενδύσεων, να πούμε και από πού τα πήραμε αυτά. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες υποδομές που δεν παράγουν κέρδος. Γιατί στο ΕΦΣΥ ε, είναι δάνειο, ε, είναι εκμετάλλευση και από την εκμετάλλευση θα πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο, δηλαδή θα πρέπει να σου αποφέρει η επένδυση. Και έχουμε 10 χιλιόμετρα ή 100 χιλιόμετρα σιδηρόδρομο που δεν ε, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΦΣΙ αλλά πρέπει να πάρει επιδότηση, όχι δάνειο. Και ε, παρακαλώ τον Επίτροπο, ωραίο είναι το blending, η ανάμειξη αυτή, αλλά ε, παρακαλώ μην τα φορτώνετε όλες τις μεταφορές. Ε, ε, θα πρέπει να παραμείνουμε στην επιδότηση λοιπόν, γιατί δεν μπορούν όλοι να πάρουν δάνεια για υποδομές. Ε, για τη σχέση μας τώρα με το δημόσιο χρέος και τη Eurostat. Στη Λιέγη έχουμε ένα μεγάλο έργο για ένα καινούριο μετρό το οποίο δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Για ποιο λόγο, διότι υπάρχει λέει δημόσιο χρέο. και προσμετράτε εκεί και αυξάνεται το χρέο. Λύνεται, έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί αν δανειστεί μια πόλη, το συνυπολογίζουν στο χρέο το κρατικό και καταλαβαίνουμε και ξέρουμε ότι το Βέλγιο είναι ήδη υπερχρεωμένο, οπότε δεν θέλει να συνυπολογιστεί αυτό. Για το blending τώρα, 1,1 ε, δις blending είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι αρκετό. Υποθέτω ότι εάν συνδυάσετε τους δύο πόρους σεφ και εύση και αυτό blending το λέτε, ε, ε, αλλά δεν χρειάζεται να παραμείνετε στο ένα δισεκατομμύριο, μπορούν ε, να σημαίνουν blending και το σεφ μαζί με το εύση. Ελπίζω να τα κατάλαβα καλά. Μετά, ποιο είναι το κράτος μέλος που λείπει, 27 μας είπατε, ποιο είναι το 28 πολύ ενδιαφέρον να το μάθουμε, ποιο δεν συμμετέχει. Αν είναι η Μεγάλη Βρετανία, τότε λύνεται το πρόβλημα. Αν δεν είναι η Μεγάλη Βρετανία, τότε τι γίνεται. Ωραία ερώτηση, δεν είναι αυτή. Έρχομαι και σε σοβαρέ ερωτήσει. Α, δεν βλέπω το χρονό. Α, το βλέπω. Ζητώ συγγνώμη, τελειώνω. Λοιπόν, ε, το Brexit τώρα τι θα σημάνει για εσά. Καλά, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μου το απαντήσει τώρα ο Επίτροπο, αλλά αν στην Ισπανία, α πούμε, φεύγει ένα πρόγραμμα, δεν εγκρίνεται και πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα έχω πρόβλημα εγώ τότε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο Ρόμπερτ Ζήλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρε, για την ομιλία σα. Ακούγεται σαν παραμύθι αυτό που είπατε και καταλαβαίνω πλήρω τι ευθύνε σα. Δουλειά σα είναι στην Επιτροπή και πρέπει να την κάνετε. Όμω, να κάνω και εγώ κάποιε κριτικέ επικριτικές παρατηρήσεις για το πώ λειτουργεί το ΕΦΣΙ. Τρία σημεία βασικά. Πρώτα απ' όλα για τη γεωγραφική κατανομή. Η έκθεση τη ΕΤΕ καταλήγει στο ίδιο. Μιλάμε για ιδιωτικό χρήμα όπου βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα υπολογίζει κανείς να έχει κέρδο. Λογικό είναι. Αυτό θέλουμε στι χώρε που υπάρχει ΑΕΠ, ε, θέλουμε βελτίωση του δικτύου μεταφορών λόγου χάρη. Δεν μπορούν όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά τα έργα δεν πηγαίνουν στην περιφέρεια τη Ευρώπη, όπου υπάρχει λιγότερη ανάπτυξη σε κάθε περίπτωση. Δεύτερο σημείο. Υπάρχουν τομεί πολιτική συγκοινωνιών, οι οποίε βρίσκονται στο σύστημα εδώ και πολλά χρόνια με τη διευκόλυνση για τη διασύνδεση τη Ευρώπη, το ΣΕΦ, με την πρόβλεψη έργων που μπορεί να μην έχουν τεράστιο κέρδος, ε, αλλά υπάρχουν διαφορετικοί πολιτικοί στόχοι εδώ, γι' αυτό υπάρχει και η κατανομή σε τομεί. Υπάρχουν πράγματα τα οποία προχωρούν καλύτερα από άλλα Πρέπει να κοιτάξουμε να έχουμε κάποιο είδου μετατόπιση. Όχι μόνο δηλαδή να γίνει καλύτερα η κατανομή των έργων, αλλά και μεταξύ των τρόπων μεταφορών και συγκοινωνιών. Και μετά για τους ιδιωτικούς εταίρους μας. Είδα τι γίνεται στην ε, Λετωνία και φαντάζομαι ότι το έχετε υπολογίσει και υποτίθεται ότι είναι ήδη στα έργα η Λετωνία. Μόλι πριν λίγε εβδομάδε υπογράφτηκε η πρώτη συμφωνία και δεν έχει προχωρήσει καν. Εάν αναλύσει κανεί αυτό είναι ένα καλό λετωνικό παράδειγμα, για τα προγράμματα μεταφορών για, την, ε, για το Δήμο τη Ρήγα, τη πρωτεύουσα. Εδώ υπάρχει ένα σκέλο για τι υποδομέ και ένα για την ανάπτυξη του τραμ. Ε, όμως το θέμα είναι ότι κανείς στο κοινό δεν γνωρίζει ποιο μέρος της επένδυσης αναλαμβάνει ποιος και σε ποιο μέρος του σκέλους του έργου αντιστοιχεί. Δηλαδή όταν ε, υπάρχει ειδικό σχεδιασμός και υπάρχει ήδη γραμμή του Τραμπ που έχει σχεδιαστεί αλλά έχει πάρει ένα ειδικό όνομα, δεν φαίνεται να πείθει αυτού του είδους ο προγραμματισμός. Μας λένε μάλιστα ότι θα περάσουμε από εκεί, από τον Εκοταφείο, ε, γιατί μας το ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά είναι σημαντικά για την άποψη του χρέους. Ο Δήμος θα αναγκάσει την εταιρεία αυτή, την ιδιωτική του Δήμου που, ε, με την οποία συνεργάζεται, να αναλάβει το παθητικό, το χρέος αυτό θα είναι επιπλέον φορτό για μα τα επόμενα 50, 15 μάλλον χρόνια. Δεν είναι διαφανή ο τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και είναι αντικείμενο διαχείριση τα έργα. Πρέπει λοιπόν να το φροντίσουμε αυτό οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε ε, που ήρθατε και στην Επιτροπή μα και για αυτά που μα είπατε. Και βέβαια το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα έρθετε εδώ να το υπερασπιστείτε. Στην Επιτροπή Μεταφορών δεν είναι τόσο εύκολο αυτό γιατί εμεί βλέπουμε ότι μα παίρνετε λεφτά το σεφ ε, και μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε με μεγάλη επιτυχία στις μεταφορές που τα χρειαζόμαστε κιόλα. Και ε, τα αηφόρα και βιώσιμα προγράμματα μεταφορών από το ΕΦΣΙ δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι ελκυστικές οι επενδύσεις, δεν προσελκύονται ιδιώτες επενδυτές. Είχαμε μια πιλωτική ε, φάση για να βγάλουμε, θυμάστε, τα λεγόμενα ομόλογα έργου τότε, για να ε, αυγατήσουν κάπως τα λεφτά. Ε, στις οδικές μεταφορές μπορεί να γίνει αυτό και βρίσκεται επενδυτές. Στην Ασία είπατε ότι υπάρχουν επενδυτές επενδυτές που έχουν ανακαλύψει το πόρταλ, τη δικτυακή πύλη, έχουν δεσμευτεί, είναι φόρες αυτές βιώσιμες επενδύσεις, μεταφορές. Και δεύτερον, ε, είπατε θέλετε να σας βοηθήσουμε, με χαρά να σας βοηθήσουμε και σε εκλογικές περιφέρειες να υποβάλουν αίτηση τα σωστά έργα. Γιατί έχετε υπόψη σας τι έργα πρέπει να είναι αυτά. Εγώ είμαι Γερμανίδα και γνωρίζω ε, και σε άλλα κράτη υπάρχει αυτό. Υπάρχουν ε, προβλήματα με την εσωτερική ναυσιπλοεία. Δεν υποβάλλονται έργα. Ε, για το σιδηρόδρομο επίσης, δεν ξέρω. Το, αυτό που ενδιαφέρει το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι οι αυτοκινητόδρομοι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, τους χρειαζόμαστε και αυτού, Αλλά βιώσιμο σημαίνει ε, ε, πλωτά ποτάμια, σημαίνει σιδηρόδρομο Τι να κάνουμε εμεί για να υποβάλλουν αιτήσει ενδιαφερόμενοι και να προωθήσουμε αυτό που θέλετε. Ορίστε, μου περσεύει και ένα λεπτό, θα το δώσω στον Ντομινίκ Ρικέ που είναι αρμόδιος για τα θέματα τα οικονομικά δικός μας. Ε, περιμένετε, χρειάζεται και δική μου έγκριση. Τι είναι αυτά, η κυρία Κίλωνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρε Κατάινεν. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε την ανάγκη να πραγματοποιήσουμε ένα άλμα και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Πρέπει το σύστημα συγκοινωνιών μα να φτάσει στα ύψη τη συμφωνία του ε, Παρισιού. Μηδενικέ εκπομπέ είναι ένα πολύ δύσκολο στόχο. Όμω έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα, είναι σίγουρο, ιδίω σε ό,τι αφορά τι οδικέ μεταφορέ. Χαίρομαι λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχει λάβει ήδη αυτά υπόψη τη, όμω ακόμη πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι τα έργα που ω τώρα έχουν περάσει από το ΕΦΣΥ μόνο κατά ένα 6% αφορούν το συγκεκριμένο τομέα. κατά έναν. η ερώτησή μου λοιπόν είναι κατά πόσον μπορούμε να κατευθύνουμε το ΕΦΣΥ και τη χρήση του προς τα έργα που θα μειώσουν, θα περιορίσουν τις εκπομπές από τις μεταφορές. Ε, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να πετύχουν ε, πιο εύκολα τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Με σαφείς προϋποθέσεις για την ε, σωστή επιλογή των έργων. Ελπίζω έμφαση να δοθεί στην ανανέωση ε, και την απόσυρση των παλαιών οχημάτων, στην ενίσχυση των υποδομών και στο να έχουμε έργα τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες μας για γενετικότητα και ελευθερότερη κυκλοφορία. Για την ώρα αυτό δεν συμβαίνει. Ευχαριστούμε κυρία Ντελή. Κύριε Κατάινεν, ε, Χαίρετε. Η προσέγγιση αυτή που έχει επικρατήσει μας ικανοποιεί. Η προσέγγιση της ΕΤΕ συμφωνεί με τους πρασίνους και τις δικές μας απόψεις. Όμως εδώ και ένα μισή χρόνο έχουν λέξει τα πράγματα με τον αδρόμο του Όσλο και της Κοπεχάγης που δεν είναι και από τις φτωχότερες περιοχές της Ένωσης και επειδή η αεροπλοεία είναι υπεύθυνη για 10% ε, των ε, συνολικών εκπομπών και 18% των ε, εκπομπών από, την, από τις αερομεταφορές και με τους στόχους του Μόντρεαλ όπως αποφασίστηκαν στο ΜΚΑΟ όλα αυτά είναι ασύμβατα με τη συμφωνία και της COP21 των Παρισίων δηλαδή και με όσα έχουμε πει ως τώρα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι απλούστατη πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, δικαιολογήσει την πολιτική εξάπλωσης και διεύρυνση των αεροδρομίων βάσει των στόχων που έχουμε θέσει για το 2030. Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Δεύτερη, ακόμη απλούστερη. Το έθιξαν και οι συνάδελφοι. Κοιτάζω τα πρώτα έργα του ΕΦΣΥ που επελέγησαν και, και παρατηρώ ότι στα τρία που επέλεξε η ΕΤΕ είναι έργα επέκταση αυτοκινητοδρόμων, Σλοβακία, Ιταλία και Γαλλία. Εάν τα κάτι μελη Εγώ νομίζω ότι το ΙΕΤΕ δεν παίζει το παιχνίδι δίκαια. Διότι είχαμε πει να μην δοθεί η μεγαλύτερη έμφαση στις οδικές μεταφορές, θέλαμε ευφυείς επενδύσεις προς τους σιδηροδρόμους, προς τις πλωτές μεταφορές, ώστε να ενισχύσουμε το συνδυασμό πολλών τρόπων μεταφορών, ε, διασυνοριακά με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τι νέε τεχνολογίε με την αξιοποίησή του. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι απλούστατη. Ακόμη και αν η κυρία Μπούλτ θύμισε ότι τα έργα που επελέγησαν θα πρέπει να είναι βιώσιμα, από την άλλη να ρωτήσω το εξή απλό. Η Επιτροπή θα ζητήσει από την ΕΤΕ επιτέλους να επιλέγει έργα τα οποία να συνάδουν με την εντολή που της δόθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάρκο Πίπε, τώρα περνάει στο μονόλεπτο χρόνο αγόρευσης. Ευχαριστώ. Και μισό λεπτό μου έχει δώσει ο Βιμ Κάμπ. Αλλά θα είμαι σύντομος. Ενάμεση έχω τώρα. Ωραία. Τώρα πέρασε το μισό λεπτό. Ήδη. Ε, ε, είναι καλά τα προγράμματα και τα έργα που έχουν ξεκινήσει. Ωραία. Υπάρχει διαφάνεια πολύ καλά, αλλά παραμένουν στα κράτη-μέλη διαφορές στην αποδοχή του νέου ε, αυτού εργαλείου. Σε χώρες που είναι χαμηλά τα επιτόκια δεν χρειάζεται το ΕΦΣΥ, βρίσκεται και άλλες επενδυτές και κρατικούς προϋπολογισμούς που συμφέρουν περισσότερο από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και πάλι αυτό είναι μεταφορά πιστώσεων προς τις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης, που δεν έχουμε αντίρρηση, διαπίστωση είναι αυτό μόνο. Τώρα, για την δεύτερη περίοδο του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Μας πήρατε λεφτά από το ΣΕΦ, ε, από το σιδηρόδρομο, από την εσωτερική ναυσιπλοεία παραμένουν λιγότερα. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επέστρεψαν κάποια χρήματα. Εμείς τη ζητάμε. Δεν μιλώ εξ ονόματος όλων, αλλά φαίνεται από την κατάσταση ε, στη δεύτερη περίοδο τώρα του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων να μην θίξετε καθόλου το Connecting Europe, να παραμείνει ισχυρή, να ξαναγίνει ισχυρή αυτή η διευκόλυνση. Από εκεί και πέρα να βρεθεί ένα κονδύλι που να χρηματοδοτήσει το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Μην πάτε πάλι να τα πάρετε από εκεί που τα χρειαζόμαστε τόσο επιγόντως, από το σιδηρόδρομο και τα ποτάμια. Ευχαριστώ. Η Μαρία Γραπίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που είστε εδώ. Βεβαίω, θα θέλαμε να μην έχουμε τόση πίεση χρόνου. Δεν μπορώ να προλάβω να πω όλα όσα θέλω όσα αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που μου δίνετε. Αλλά να επιστρέψω στην ομιλία σα. Είστε πολύ πιστικό. Κάθε φορά που στην Ολομέλεια μα πείθετε. Όποτε όμω βγαίνουμε στην πραγματικότητα και στην πραγματική ζωή, στι εκλογικέ μα περιφέρειες, βλέπουμε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Και εγώ ακολούθησα τη συμβουλή σα, Πήγα στου ψηφοφόρου μου και του ρώτησα πώ ε, πιστεύουν ότι μπορούμε καλύτερα να αξιοποιήσουμε το ΕΦΣΥ. Τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα. Πρόσφατα συμμετείχα σε μια διασυνοριακή διάσκεψη με εκπροσώπους από τοπικές κυβερνήσεις, δημάρχους, από χωριά και κομοπόλεις και πολύχνης στα βουνά με τεράστια προβλήματα ε, υποδομών. Πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται με τη σωστή κατανομή, τη γεωγραφική κατανομή, ιδίως με τις στοχότερες περιοχές το ΕΦΣΥ υποτίθεται ότι θα προωθούσε την ανάπτυξη. Αν δεν πάνε κονδύλια ως εκεί, πώς θα τους βοηθήσουμε. Τι γίνεται με αυτά τα κριτήρια. Δεν μπορεί να ισχύει μόνο το όποιο φτάσει πρώτος ε, πρόλαβε. Ε, πρέπει να έχετε λίγο πιο αυστηρό κριτήρια επιλογή. Η χρηματοδότηση έχει μεγάλο αντίκτυπο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Στην ε, περιφέρεια τη Μισοάρα, υπήρχε μια ε, εκπρόσωπο τη Βουλγαρία, ήρθε μια εκπρόσωπο τη Βουλγαρία που μας μίλησε για το πρόβλημα της παλαιότητας του στόλου και έχουν μεγάλη δυσκολία με την απόσταση και την ανανέωση των σκαφών τους. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό ας πούμε. Ευχαριστώ πολύ, Ντομινίκη, και ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, που ήρθατε πολύ σύντομα. Πρώτη παρατήρηση για το FC1, ενδιάμεσο απολογισμό κάνουμε. Θυμίζω στα ποσοτικά στοιχεία ότι 30% ε, υποτίθεται θα πήγαινε στις μεταφορές. Ε, και 75% ε, επενδύσεις για το FC1, ενώ είμαστε στα 11 δις και 138 είναι ο συνολικός όγκος. Δηλαδή απέχουμε πάρα πολύ από το στόχο για τις μεταφορές, ενώ πήρατε πολλά λεφτά από το ΣΕΦ για το Ταμείο Εγγύησεων. Προς το παρόν είναι ένα δις και κάτι στην κινητοποίηση. Άρα, αυτά που μας πήρατε από το Connecting Europe δεν θα ε, ε, έχει την απαραίτητη μόχλευση για το FC1. Είναι λιματική για τις μεταφορές αυτή η συναλλαγή. Δεν θα μιλήσω για τα γεωγραφικά, για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τα οριζόντια έργα, Εντάξει, γενικά είναι σωστά. Για το blending τώρα. Δηλαδή να υπάρχει ένα συνδυασμό επιδοτήσεων και δανείων. Έτσι, το χρηματοδοτικό μέσο που λέγεται ΕΦΣΙ. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και πρέπει, κύριε Επίτροπε, να γίνει ένα συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Δηλαδή, να μην είναι ξεκάρφωτα αυτά και άσχετα μεταξύ τους με την Τράπεζα Επενδύσεων και το blending να αφορά και τα έργα. Δηλαδή, μιλήσατε προηγουμένως αλλά και όλα αυτά που έχει αναλάβει ο εκτελεστικός οργανισμός στα ε, έργα τα οποία έχουν κατατεθεί ε, χωρίς να επιλεγούν αυτά θεωρούνται νεκρά. Όχι. Ε, να μπορούν στη συνέχεια να επανεξετάζονται. μιλήσατε για τον κανονισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι ανησυχούν πάρα πολύ. Οι Αμερικανοί πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση και σας επιτρέπ, μου επιτρέπετε να κάνω μια πρόταση για τη φερεγγιότητα των κρατών μελών, για το δημόσιο χρέος και την αδυναμία ε, να δράσουν εντός του Συμφώνου Σταθερότητας. Αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει να συνυπολογίζονται ε, με βάση την απόσβεση του έργου ε, και να μην υπολογίζεται απλώς μηχανιστικά ε, σε δύο χρόνια στο δημοσιοχρέο. Εδώ πρόκειται για έργα μακρά πνοή για 40 χρόνια. Θα πρέπει να υπολογίζουμε την απόσβεση και το κέρδο σε ορίζοντα 30 ε, ετία. Για το f 2 λοιπόν. Συμφωνούν και οι συνάδελφοι του ΕΛΚ. Ε, δεν θα πρέπει να πάρουμε λεφτά από το ΣΕΦ, μάλλον να βάλουμε ξανά περισσότερο για να αυξηθεί η προοικοδότηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Βόζεμερκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Πίτροπε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας κάνατε. Θέλω να σας ρωτήσω, εν γνώση ότι το επενδυτικό πακέτο, πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να το προβάλλουμε, στην Ελλάδα έχει προβληθεί, ήδη επισημάνατε μια επισκεψιμότητα που παρουσιάζεται στο πόρταλ. Θέλω να επισημάνω με αφορμή την, το επενδυτικό, την επενδυτική πλατφόρμα Energy Positive που έχει χαρακτηριστεί ότι εντάσσεται στο success story αυτής της επενδυτικής πολιτικής. Και είναι γνωστό ότι εφαρμόζεται στο Παρίσι για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων με ε, τουλάχιστον ε, 11 δημοσίου τομεί, έτσι δεν είναι, και δύο χρηματοδοτικού φορεί και δύο ιδιωτικού φορεί. Θέλω να σα ρωτήσω εάν μέσω αυτή τη επενδυτική πλατφόρμα στην Ελλάδα θα μπορούσε η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί αυτή την πλατφόρμα και να ε, μπορέσει να εκμεταλλευτεί ε, τις ευκαιρίες του επενδυτικού σχεδίου αυτού για τον τομέα των μεταφορών και, του τουρισμού που είναι ουσιαστικά για τη δική μου τη χώρα η βασική στρατηγική τομής, ιδιαίτερα στην οικονομική θέση που βρίσκεται τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ινέσα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι κάπως έκπληκτη εδώ γιατί ε, ε, νομίζω ότι πρόκειται να μου κάνετε κάποιο δώρο, κάποια επιπλέον λεπτά και τελικά μάλλον δεν θα γίνει. Λοιπόν, εγώ ήδη ε, έχω καλέσει εδώ τι επιχειρηματίε από την περιοχή μου για να μας το εξηγήσει το πακέτο Juncker. Ε, έχει πάει και η ΕΤΕ εκεί για να τους κάνει κάποιες παρουσιάσεις. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ενημέρωση. Και εμείς έχουμε διδαχθεί πολλά και εσείς για το ΕΦΣΙ και για το 1 και για το 2. Αυτό που έχουμε καταλάβει λοιπόν είναι το εξή. Αν στο ΕΦΣΙ 1,0 είχαμε το εξή αποτέλεσμα 25% του ΣΕΦ να εξαφανίστηκε, τελικά διαπιστώσαμε ότι μόνο 8% ήταν η απόδοση για εμάς. Ενώ για την ενέργεια, για παράδειγμα, η ουσιαστικά εκεί ήταν το 25%. Άρα λοιπόν είπαμε ότι εμείς από τις μεταφορές βάζουμε ποσά στο ΕΦΣΙ και τα χρησιμοποιούν για δικό τους πλεονέκτημα στην ενέργεια και σε άλλους χώρους. Φοβάμαι λοιπόν ότι με το ΕΦΣΙ 2,0 ε, θα συμβεί το ίδιο. Ή λοιπόν θα περιχαρακώσουμε τα ποσά και θα πούμε ότι βγάζουμε από το ΣΕΦ εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε στο, για μας στις μεταφορές ή να προσέξουμε πιο πολύ, να έχουμε λοιπόν ε, κάποιες ε, προσπάθειες, για παράδειγμα μείωση των εγγυήσεων, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με καλύτερο τρόπο για τα δικά μας θέματα. Επίση, αν διατηρήσουμε τα κονδύλια αυτά στο Connecting Group Facility, θα μπορούσαμε αυτό το, αυτή την ανάμεξη να την κάνουμε εμεί με την ΕΤΕ, γιατί διαφορετικά εξαφανίζονται τα κονδύλια, φεύγουν από τι μεταφορέ και δεν ξέρουμε πού καταλήγουμε. Αυτά ζητήσαμε και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ότι εσεί το θέμα των αυτοκινητοδρόμων το αφαιρέσατε. Γιατί ναι, εντάξει, δεν είναι ότι πιο βιώσιμο, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να διατηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε αυτέ τι υποδομέ τι οποίε χρειάζεται με δραματικό τρόπο η Ευρώπη. Τουλάχιστον λοιπόν θα έπρεπε να μπορούν να διατηρηθούν αυτά μέσα στο ΕΦΣΥ. Ευχαριστώ πολύ Ινές. Είπα στην αρχή οι συντονιστές έχουν περισσότερο χρόνο και μετά ο καθένας ένα λεπτό. Και εσύ ε, ζήτησε το λόγο πολύ αργά, γι' αυτό ε, στο δώσαμε και αργά. Δεν είπα αυτό, λέει ότι είμαι εισηγήτρια και είχα παραπάνω χρόνο κανονικά, δεν πειράζει. Ο κύριος Ντελή. Oh, Μπορώ. Μάλιστα. Ουσιαστικά, Καταρχά σα ευχαριστώ που ήρθατε. Και δύο-τρία πραγματάκια να πω κι εγώ. Πρώτον, την τελευταία φορά ε, που μπήκα στο site της ε, Τράπεζας Επενδύσεων είδα γύρω στα 89 έργα, κάτι τέτοιο πολύ εντυπωσιακά. Αλλά μας λέτε μόνο 16 είναι των μεταφορών. Εντάξει, άμα το δεις είναι χαμηλό ποσοστό αυτό. Και κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν και σε αυτό και ανησυχούν για την γεωγραφική ε, κατανομή που είναι δυσανάλογη. Τρία έργα είναι από ε, την ε, περιφέρεια της Κεντρικής Ευρώπης και ένα συνδέεται με τις μεταφορές. Εν πάση περιπτώσει. Μιλήσατε για ξένους επενδυτές. Εξ όσων γνωρίζω, αυτοί οι ξένοι μπαίνουν σε πλατφόρμες. Δεν ε, χρηματοδοτούν το έργο αυτό καθ' αυτό. Διορθώστε με αν ασφαλώ. Ε, τι γίνεται αν θέλει ένας Ασιάτης επενδυτής να έρθει να επενδύσει σε ένα από αυτά τα έργα ή τις πλατφόρμες. Πώς έχει η τι πλατφορμες Υπάρχει ήδη κινέζικη ηδη αραβική παρουσία, φερρυπίν. Θα με ενδιέφερε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ακριβώς αυτό ήθελα και εγώ να ρωτήσω, αυτό που ο κύριος Δέλη για τι οικονομικέ επενδύσει. Την ε, χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό ιδιωτικό τομέα ε, για το ΕΦΣΥ. Μπορείτε να σχολιάσετε και να μα πείτε πώ έχουν αλλάξει οι μορφέ χρηματοδότηση μετά από αυτό που έγινε στις ΗΠΑ, το αποτέλεσμα των εκλογών, τι ρατραχέ τη αγορέ, το Brexit, όσα συμβαίνουν εκτό Ευρώπη τέλο πάντων και το πώ επηρεάζονται οι αγορέ. Θα ήθελα λοιπόν τι δικέ σα ε, παρατηρήσει μετά την πείρα που έχετε συγκεντρώσει στον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μοντέιρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ να χαιρετήσω την παρουσία εδώ του Αντιπροέδρου Κατάιναν και εντάχει να πω ότι η Επιτροπή αυτή είναι Επιτροπή Μεταφορών αλλά και Τουρισμού. Και επειδή μιλάμε για ένα κλάδο με ιδιαίτερο βάρος για, οικονομία, για τις οικονομίες των χωρών μας, αλλά και τη Ευρώπη συνολικότερα, ήθελα να ρωτήσω συγκεκριμένα. Γνωρίζετε τι έργα προέκυψαν στον τομέα του τουρισμού και έχουν ε, καλυφθεί από το ΕΦΣΥ. διότι μας ενδιαφέρει τι θα γίνει και σε επίπεδο χωρών. Εγώ ως Πορτογαλίδα οργανώνω μια πλατφόρμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Θέλουμε λοιπόν να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο μπορούν να βρεθούν κονδύλια μέσω από αυτό το πρόγραμμα. Τι συμβουλές μας δίνετε και πώς μπορούμε να εργαστούμε από κοινό ώστε αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξελιχθούν καλύτερα, ώστε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το τόσο σημαντικό ταμείο για να δημιουργηθούν ε, περαιτέρω θέσει απασχόληση. Ευχαριστώ. Σας Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Θα γνωρίζετε ε, το έργο Vanguard που συμμετέχουν διάφορες περιφέρειες. Εχθές συνεδρίασαν εδώ στο Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά έχουν το εξής πρόβλημα. Συνεργάστηκαν διάφορες περιφέρειες τα γνωρίζετε αυτά πολύ χρόνο τώρα. Έχουν πιλωτικά προγράμματα που απευθύνονται στην ε, βιομηχάνηση 4,0, στην τεχνολογία. Όταν όμως χρειάζεται να κάνουν την ανάπτυξη και τις εφαρμογές για συγκεκριμένα προϊόντα έχουν πρόβλημα. Δεν είναι επιλέξιμα ούτε για το Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων, ούτε για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δεν είναι επιλέξιμα για καμία χρηματοδότηση. Ενώ πρόκειται για την εχμή της τεχνολογίας και ε, για αυτά τα πράγματα μιλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς σκέφτεστε να υπάρξει καμία ευελιξία εκεί στο σχέδιο Juncker ή δεν ξέρω σε κάποιο άλλο πρόγραμμα για να χωράνε και οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν ε, καταφέρει ε, τεχνολογική συνεργασία με πανεπιστήμια, με ιδρύματα, με ε, βιομηχανίες και εταιρείες εχμής οι που συμμετέχουν. Εδώ σας ανακοινώνω, θα το ξέρετε και σας έχουν διαβιβάσει και το γνωρίζω το εξή. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λάβει μια σημαντική απόφαση για να τους βοηθήσει, ενδέχεται όλη αυτή η δουλειά να πάει στο βρόντο. Οπότε αυτό αποθαρρύνει, καταλαβαίνετε, και τις εταιρείες και τα τεχνολογικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια που τόσο καιρό κοπιάζουν και συνεργάζονται και δίνουν και σημασία στα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε για τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, το ΣΕΦ. Είναι θαυμάσια τα έργα και όταν μας λέτε ότι έχουμε τόσα λεφτά κερδίσει, αλλά τι γίνεται με τα έργα. Τα έργα πάνε στην άλλη κατεύθυνση από αυτά που μας ενδιαφέραν. Γιατί θέλετε να σταματήσετε την κλιματική αλλαγή, να ενώσετε την Ευρώπη και να δημιουργήσετε δουλειέ. Όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στα έργα που εγκρίνεται. Παράδειγμα. Βαλανσιέν Βρυξέλλες, το τρένο. Λείπουν 800 μέτρα σιδηρόδρομο, ράγα κανονικά θα ε, κερδίζαμε ένα χρόνο ε, μια ώρα στη διαδρομή Βρυξέλλε Βαλανσιέν με το τρένο. Πώ θα το λύσετε αυτό. Ή Βερολίνο Βρότσλαβ. Λείπουν 50 χιλιόμετρα. Ε, θα μπορούσαμε 100 εκατομμύρια να γλιτώσουμε και δύο ώρες ή αντίστοιχα ε, γύρω από το Βερολίνο. Λείπει μια γέφυρα. Πάλι 100 εκατομμύρια θα μπορούσαμε να κερδίσουμε 2 ώρε και 40-50% μεταφορά από τον αυτοκινητοδρόμο στο σιδηρόδρομο. Αυτά ε, είναι και οικολογικά. Εσείς πώς επηρεάζετε τα έργα ώστε να στρέφονται στη σωστή κατεύθυνση και τους στόχους τους δικούς σας, τους εκπεφρασμένους. Και ο κατάλογος θα μας τον δώσετε των εγκεκριμένων προγραμμάτων και εκείνων που σχεδιάζετε, που προγραμματίζετε και για ποιο λόγο χρηματοδοτείτε ένα πρόγραμμα, επιλέγετε ή ε, απορρίπτετε. Ξέρω ότι σας πιέζει ο χρόνος, αλλά τώρα μπορείτε και να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Φεύγω για την Ινδία και έχω πέντε λεπτά στη διάθεσή μου. Θα προσπαθήσω να είμαι συνθετικός. Όλα τα έργα τα οποία έχουν υπογραφεί θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ, γιατί ενημερώνεται πρόσφατα και κάθε φορά που γίνεται κάποια πράξη. Γιατί έχουν επιλεγεί αυτά. Στο FC 2,4 υπάρχει μια εφαρμογή που εξηγεί για ποιο λόγο έχουν επιλεγεί και αυτό είναι μια από τις αλλαγές που φέραμε. Γιατί θέλουμε να μπορούν όλοι να διαπιστώνουν την ε, προστιθέμενη αξία του ΕΦΣΙ, κάνοντας αυτές τις συγκρίσεις ε, με τα όσα τρέχουν με τις άλλες διαδικασίες. Όχι άλλες περικοπές. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε άλλο κονδύλι από το Connecting Europe. Αντίθετα, ε, οι επιχορηγήσεις του Connecting Europe θα αυξηθούν κατά 1,1 δις. Και αυτά για την ανάμεξη, για αυτό το χαρμάνι που κάνουμε. Άρα 1,1 δις σε χορηγήσεις με αποτέλεσμα η επίπτωση του ΕΦΣΙ να μεγιστοποιείται, γιατί μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει έτσι project τα οποία δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει κανείς μόνο από το ΕΦΣΙ, είτε γιατί οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές, είτε για κάποιο άλλο λόγο. Άρα λοιπόν είναι τελείως νέο προϊόν. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλή συμφωνία. Δεύτερον, το ΕΦΣΙ 2,0 λέει στον κανονισμό πως τουλάχιστον 40% της χρηματοδότησης του ΕΦΣΙ θα πρέπει να δοθεί στους στόχους του COP21, της COP21, το οποίο σημαίνει πολλά και διάφορα. Μπορεί να είναι μεταφορές, μπορεί να είναι ενέργεια, μπορεί να είναι εξοικονόμηση ενέργειας κτλ. Γεωγραφική κατανομή. Πρόκληση όντως. Καμιά φορά είναι σαν να σπρώχνουμε, να σπρώχνουμε και να μην μετακινείται τίποτα. Σε κάποια κράτη υπάρχει τόσος δισταγμός. Και είναι εντυπωσιακό. Υπάρχουν και πολιτιστικοί λόγοι που διστάζουν κυβερνήσεις και επιχειρήσεις και υπάρχουν και διαφορές μέσα σε γειτονικές χώρες, για παράδειγμα. Στη... Κοιτάξτε τη Βουλγαρία. Τρεις τράπεζες έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες χρηματοδότησης με τον ΕΦΣΙ, δηλαδή ε, χρηματοδότηση των μικρομεσών επιχειρήσεων τη Βουλγαρία. Εγώ πήγα στη Ρουμανία. Είδα τους τέσσερις διευθύνοντες συμβούλους των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών και μας είπαν δεν χρειάζεται, δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό. Στη Ρουμανία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν παίρνουν δάνεια γιατί οι τράπεζες λένε ότι δεν υπάρχει ζήτηση και μας δεν μας ενδιαφέρει. Δεν τους καταλαβαίνω. Ίσως υπάρχει κάποια λογική πίσω από αυτό, αλλά εγώ δεν τη βρήκα. Τώρα σε κάποιες χώρες η κεντρική κυβέρνηση όταν τους εξηγώ τι είναι το FC, μας λένε ωραία, ωραία. Δεν είναι χορηγία, δεν είναι δάνειο. Α, τι είναι ακριβώς χρηματοδοτικό εργαλείο. Α, δεν μας ενδιαφέρει. Ενώ κάποιες από τις περιφέρειες είναι πιο προχωρημένες στον τρόπο που σκέπτονται. Και πολλές φορές εγώ ενδιαφέρομαι περισσότερο στο να συναντήσω τις ηγεσίε των περιφερειών παρά τις κυβερνήσεις. Γιατί πολλές φορές η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση και οι δήμαρχοι είναι πολύ πιο ανοιχτοί στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις στα smart cities, δηλαδή ευφυείς πόλεις, ψηφιακή επένδυση, ε, πολλές φορές ευφυείς μεταφορές και συγκοινωνίες. Είναι εξαιρετικοί οι δήμαρχοι, πολλές φορές είναι και ιδιαίτερα διεθνείς και κοιτάνε να δουν τι ευκαιρίες υπάρχουν. Για παράδειγμα, όταν προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε πως η ευκαιρία του να συνδυάσει κανείς διαφορετικά ταμεία με Connecting Europe και ΕΦΣΥ, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες ε, πρέπει να σας πω, είναι πιο μπροστά από ό,τι κυβερνήσεις. Και γι' αυτό έχω επαναλάβει χιλιάδες φορές πως χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια να περάσει το μήνυμα. Όχι μόνο στους υπουργού, στις ηγεσίες των περιφερειών και στον ιδιωτικό κλάδο. Τι ευκαιρίες υπάρχουν και να τους δείξουμε το website για να πάρουν από εκεί πληροφορίες. Και καλά παραδείγματα. Τι κάνουν οι υπόλοιπε χώρες, τι κάνουν οι άλλες περιφέρειες, πώς τα χρησιμοποίησαν. Τώρα για το θέμα της Ελλάδος και για την πλατφόρμα, να σας πω πως ένα από τα έργα τα οποία θέλω να σας παροτρύνω να κοιτάξετε είναι αυτό της εξοικονόμησης ενέργειας που γίνεται στο Ile de France, στην περιοχή του Παρισιού, όπου, όπου έχουν ένα ΣΔΙΤ, εταιρεία ΣΔΙΤ δηλαδή, που συλλέγει 40.000 ε, κτίρια για να κάνουν ενεργειακή αναβάθμιση ε, του κτιρίου. 40.000 διαμερίσματα με συγχωρείτε και η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι 80 ευρώ το μήνα ανά νοικοκυριό. Δηλαδή 40.000 διαμερίσματα και μερική χρηματοδότηση από το ΕΦΣΥ με τεχνική βοήθεια από την πλατφόρμα. Οπότε το ίδιο μοντέλο θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα ή στην Πορτογαλία στον κλάδο του τουρισμού για παράδειγμα. Δηλαδή στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία όπου οι τράπεζες δεν έχουν την δυνατότητα χρηματοδότησης που θα ήθελαν ή που οι επιχειρηματίες δεν βρίσκουν δάνεια. Αυτή είναι η περίπτωση της Ελλάδος. Εάν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ΣΔΙΤ με μια πλατφόρμα που θα συλλέξει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πει ας πούμε ε, μικρά ξενοδοχεία ή κάποιο άλλο είδους επένδυση. Μπορεί τα κεφάλαια να τα βάλει και τα μακροπρόσωμα δάνεια του ΕΦΣΥ. Και θα μπορούσε η κυβέρνηση, για παράδειγμα, να βάλει και ποσά ω μετοχικό κεφάλαιο από τα διαφορετικά ταμεία. Και εκεί να μπει και ο ιδιωτικό κλάδο. Έτσι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να παρακάψουν το τραπεζικό πρόβλημα και να βρουν χρηματοδότηση για την επένδυση από εκεί. Όμως, καμιά φορά, στην περίπτωση τη Ελλάδα πάλι, ο υπουργό ο οποίο είναι υπεύθυνο για τα διορθωτικά ταμεία, ξέρει. Τα ξέρει και έχουμε συνεργαστεί μαζί του. Ο Μιγγέλ έχει πάει στην Αθήνα πολλές φορές. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και ελπίζω πως κάποια αποτελέσματα θα δούμε. Όμως σε γενικές γραμμές, καμιά φορά αντιμετωπίζουμε δυσκολίες όταν οι κυβερνήσεις μας λένε πως δεν μας ενδιαφέρουν ιδιωτικέ επενδύσεις. Μόνο δημόσιες επενδύσεις μας ενδιαφέρουν. Γιατί τότε δείχνουμε στους ψηφοφόρους μας ότι εμείς τα καταφέραμε. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τι μας λένε. Και γι' αυτό θα πρέπει να παρακάμψουμε αυτά τα προφανή προβλήματα. Εσείς ξέρετε την εκλογική σας περιφέρεια, εσείς ξέρετε τους περιφερειακούς ε, άρχοντες, εσείς ξέρετε τις εταιρείες που έχετε πρέπει να είναι πιο ενήμεροι. Και ένα πιο συγκεκριμένο θέμα για το τι μπορείτε να κάνετε, αν το θέλετε, είναι να οργανώσετε εκδηλώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τουριστικό κλάδο, για παράδειγμα, ή σε οποιοδήποτε κλάδο, που να πάνε οι περιφερειακοί άρχοντες και να ε, καλέσετε εκπροσώπους της Κομισιόν να τους, παρουσιάσουν το ΕΦΣΥ και από την ΕΤΕ μπορείτε να καλέσετε κάποιους εκπροσώπους, να τους πούνε τι έκανε το ΕΦΣΙ και να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα. Αυτές οι δύο λοιπόν ε, ε, ε, οι δυνατότητες εκπροσώπησης είναι στη διάθεσή σας. Οργανωθείτε, κάντε εκδηλώσεις, ενημερώστε. Έτσι θα χρησιμοποιήσετε πιο αποτελεσματικά το ΕΦΣΙ. Και βέβαια για τα βιώσιμα έργα, εγώ είπα πως το 2,0 στο ΕΦΣΙ 2,0 Αναφέρουμε στον κανονισμό πως τουλάχιστον 40% θα πρέπει να είναι χρηματοδότηση σε στόχους κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, συγκοινωνίες και μεταφορές με χαμηλές κομπές άνθρακα, προφανής περίπτωση. Επίσης, ε, κάποιοι σταθμοί ε, φόρτισης, που δεν είναι πολύ δημοφιλής, γιατί αυτή τη στιγμή η φόρτιση μπαταρία με αυτόν τον τρόπο δεν κρατάει πολύ χρόνο και δεν έχουμε την τεχνολογία που θα έδινε μεγαλύτερη διάρκεια φόρτισης. Οπότε αυτή τη στιγμή η απόδοση στι επενδύσει δεν είναι επαρκή σε οι εταιρείε να μπουν σε αυτό το χώρο. Εκεί το ΕΦΣΙ θα μπορούσε να το καταφέρει, κυρίω αν μιλάμε για διασυνοριακά έργα. Δηλαδή, αν θέλουμε την ηλεκτρο κίνηση, θα πρέπει αυτούς τους σταθμούς να τους έχουμε και εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ενέργεια, Βιοενέργεια, βιοκαύσιμα. Και αυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Όπως επίσης και το Smart Cities, οι έξυπνες πόλεις. Πολλοί δήμαρχοι, πολλές φορές, είπαν πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά το Εύση για τέτοιου είδους λύσεις. Και πρέπει να σας πω πως η Επίτροπος κυρία Μπούλτς πρότεινε κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις να παραγγείλουν μαζί ηλεκτρικά λεωφορεία. Και αντί να παραγγείλει 40 ή 50 η Μπρατισλάβα, να βρεθούν άλλες 5 πόλεις και να παραγγείλουν 5.000. Αυτό τι θα έκανε, θα μείωνε την τιμή απόκτηση. Και τότε το ΕΦΣΙ θα μπορούσε να δώσει κάποιο χρηματοδότηση. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να χρησιμοποιηθεί με πολύ έξυπνο τρόπο και είμαι έτοιμος να συνεργαστούμε αν θέλετε βοήθεια, αν θέλετε ενημέρωση, ελάτε σε επαφή μαζί μας, αλλά χρησιμοποιηθείτε και αυτούς που έχουμε επιτόπου. Γιατί είναι σημαντικό οι πόλεις και οι περιφερειακοί άρχοντες να κατανοήσουν πως έχουν τη δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία της Κομισιόν και της ΕΤΕ, αυτούς τους ανθρώπους που είναι παρόντος στη χώρα τους. Και Δύο σχόλια ακόμα. Το FC 2,0 ξεκάθαρα θέλουμε να πούμε πως δεν θέλουμε δεν θέλουμε άλλους αυτοκινητοδρόμους στα παλιά κράτη-μέλη που να χρηματοδοτούνται το ΕΦΣΙ, μόνο στα, στα κράτη συνοχής ή μόνο σε διασυνοριακά project μεταξύ κράτους συνοχής και άλλου κράτους μέλους. Γιατί? Οι αυτοκινητόδρομοι που χρηματοδοτούνται από το ΕΦΣΙ στη Γερμανία δεν έχουν νόημα. Αν ο αυτοκινητόδρομος δεν είναι κερδοφόρος στη Γερμανία, δηλαδή και πού θα είναι. Και γι' αυτό δεν θέλουμε άλλα τέτοια έργα. Εκτός, επαναλαμβάνω, αν εμπλέκεται κάποιο κράτος συνοχής. Επίσης, η αναβάθμιση. Αναβάθμιση, ναι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι λογικό. Αλλά ναι, αυτοκινητόδρομοι σε παλιά κράτη-μέλη ή σε πολύ αναπτυγμένες χώρες δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Οι διεθνείς επενδυτές έχουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες, γιατί από τα όσα μου λένε εμένα, αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλές οι τιμές για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη, οπότε αν επενδύσουν στις υποδομές, ακόμα και στα ακίνητα, ε, αυτό θα βοηθήσει να ανέβουν και οι τιμές. Και οι τιμές μετοχών είναι πάρα πολύ χαμηλές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Οπότε εκεί έχουμε κάποιες ε, ελπίδες πως θα αυξηθούν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι ε, ελκυστική για άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις και νομίζω ότι οι Κινέζοι επενδύουν όλο και περισσότερο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πρέπει να το δούμε. Αλλά οι επενδύσεις σε κανονικούς φυσιολογικούς κλωάδους είναι μια χαρά και καλωσορίζουμε όλοι τα κινέζικα κονδύλια αν έχουν σκοπό να φέρουν ανάκαμψη στην Ευρώπη. Βέβαια προκύπτουν κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη όλοι οι εμπλεκόμενοι και τα κρατημέλη σχετικά. Υπάρχει και η αβεβαιότητα η οποία δηλητηριάζει πάντα τις επενδύσεις και σήμερα το πρωί τα αποτελέσματα τα εκλογικά δεν διευκόλυναν την κατάσταση καθόλου. Δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει αυτό μέσω μακροπρόθεσμα. Ελπίζω όχι δραματικά. Και τέλος, ξέρατε πως το ΕΦΣΙ έχει κλείσει μια συμφωνία με 200, 220 τράπεζες εθνικές και περιφερειακές ή εθνικές τράπεζες επενδυτικές για χρηματοδότηση σε 280.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, 280.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, που θα χρηματοδοτηθούν ως αποτελέσματα αυτών των deal μεταξύ τραπεζών και εύση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι τράπεζες που δίνουν τη χρηματοδότηση εύση στους επιχειρηματίες, ποτέ δεν λένε ότι είναι κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά τα οποία δίνουν. Uh, και εμεί του παροτρύνουμε. Πείτε το. Γιατί με μεγάλη χαρά ε, δίνουν αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πιστεύω ότι θα ήταν απλώ δίκαιο να το λένε τη στιγμή που το κάνουν. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Καλή, ε, καλό ταξίδι, καλή πτήση προς το Δελχή και καλή επιτυχία. Επόμενο θέμα. Εφοδιαστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδυασμένε μεταφορέ στου νέου διαδρόμου διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Έξι πρωτοβουλίε είναι αυτή η δικιά μα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ινέσα Γιάλα Σέντερ, η οποία έχει το λόγο. Eh. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ του συναδέλφου μου για τις ε, προσπάθειές τους να καταθέσουν προτάσεις τροπολογιών για να βελτιώσουν το κείμενο. Και εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή για μια σειρά συμβιβαστικών τροπολογιών έτσι ώστε να βελτιωθεί και να εμπλουτιστεί το κείμενό μου. <laughs> Ε, η αρχική πρότασή μας δηλαδή. Θα ήθελα να σας πω ότι Θα συνεδριάσουμε με τους σκιώδεις συζητητές ε, για να προσπαθήσουμε να ε, κάνουμε συμβαστικές τροπολογίες και να τις υποβάλουμε στην Επιτροπή μας. Βέβαια, σας προειδοποιώ από τώρα ότι θα προσπαθήσω να διατηρήσω όσο γίνεται ε, μια μεγαλύτερη προβολή των εμπορευματικών μεταφορών, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, δέχτηκα κάποιες από τις προτάσεις, δηλαδή, εντάξει, να προβάλλουμε τις μεταφορές, τις εμπορευματικές, στην εφοδιαστική, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει προβλήματα με αυτά που προτείνουμε, θα πρέπει κάποιο να αναλάβει έτσι ένα συντονιστικό ρόλο να τα βλέπει εγκάρσια όλα αυτά τα θέματα. Στη συνέχεια, υπάρχει μια ανάγκη τα εθνικά προγράμματα να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τον ευρωπαϊκό προγραμματισμό, ε, αλλά και παραπάνω. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει ε, να το ζητήσουμε με τέτοιο ακραίο τρόπο, να υπάρχουν και κυρώσεις, δηλαδή να χρησιμοποιείται και το ευρωπαϊκό εξάμεινο ακριβώς ε, ως δαμόκλια σπάθη, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι σε περίπτωση που τα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα δεν συνάδουν με αυτά που ε, συμφωνούν στο Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, εναπίπτει και κάποια σχετική ράβδος. Στις συνδυασμένε μεταφορέ εσεί αναφερθήκατε και στα αεροδρόμια, ότι είναι κόμβοι, ε, εν περιπτώσει, και δίκτυα συγκοινωνιών και μεταφορών, τα λαμβάνω υπόψη. Επίση υπάρχει μια κάποια αντίσταση σε μερικές τροπολογίες που εκφράζουν επιφυλάξει ε, ως προς ε, την ε, δυνατότητα στις εμπορευματικές μεταφορές να έχουμε στα διευρωπαϊκά δίκτυα σύνδεση μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν είναι στο ε, πολιετές πρόγραμμα και στους μεγάλους διαδρόμους που έχουμε πάντα πρόβλημα ε, έλλειψης χρημάτων. Να υπάρχει αυτή η διασύνδεση και χρηματοδότηση από το ΣΕΦ τα εθνικά προγράμματα. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις Στο ΣΕΦ όμως υπάρχουν και εκεί τα δύο επίπεδα, το ετήσιο και το πολιετές. Οπότε θα προτείνω και εγώ να διατηρηθεί τουλάχιστον σε μία από τις δυνατότητες προκήρυξης αυτή η δυνατότητα. Στη συνέχεια υπάρχει όλο το θέμα που έχει να κάνει με τους κόμβους των συνδυασμένων μεταφορών και εφοδιαστικής της πόλης είναι ένα θέμα. Υπάρχει συμφωνία για τους κόμβους αυτούς και δυνατότητα ίσως και ανάγκη στο μέλλον που δεν είναι και τόσο απότερο αυτό το μέλλον, να ρυθμιστεί. Η εφοδιαστική στις πόλεις έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί εκεί πολλές φορές καταραίει ε, ο συνδυασμός των διαφόρων μεταφορικών μέσων και δεν γίνεται απρόσκοπτα η συνεργασία τους. Το άλλο θέμα, τα μέτρα και τα σταθμά. Ξέρω ότι υπάρχει εκεί πρόβλημα και επιφυλάξεις από πλευράς κάποιων συναδέλφων. Εγώ ξεκολουθώ να πιστεύω ότι εφόσον δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στη δυνατότητα να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις και να υπάρχει μια συνέχεια στα δίκτυα, αν σπάσει το σημερινό status quo των μεγάλων φορτηγών δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να προχωρήσει αυτό. Είναι και το θέμα της αυτοματοποίησης, αλλά δεν τα βλέπω όλα τόσο, με, έτσι, τόσο ρόδινα. Έχω τις επιφυλάξεις μου Συμπέρασμα. Λαμβάνω υπόψη μου όσο γίνεται περισσότερο τις τροπολογίες ε, που έχουν υποβληθεί, ιδιαίτερα τις το σκεπτικό τους και την κεντρική ιδέα για να τις συμπεριλάβω τις συμβαστικές που θα έρθουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ευχαριστώ. Η Κλάουντια Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. με λίγο γιατί 210 τροπολογίες για μια έκθεση πρωτοβουλίας που δεν είναι και επίμαχη νομίζω ότι το παρατραβάνε. Ε, υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία διαφωνούμε, έτσι σημεία τριβής Παράδειγμα, οι τροπολογίε για το διοξίδιο του άνθρακα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βεβαίως δεν είναι ε, κατά της μείωση ε, των εκπομπών των ε, βλαβερών ρήπων. Απλώς είναι πολύ ακραίες κάποιες τροπολογίες και θα πρέπει στους συμβιβασμούς να μετριαστούν και να αλλάξουν και να μπορέσουν να συμφωνήσουν όλοι. Γιατί εκτός από το περιβάλλον έχουμε και ανθρώπους και ανάγκες της οικονομίας που πρέπει να κυριαρχούν, όχι μόνο το περιβάλλον. Αυτό μόνο με συμβιβασμό μπορούμε να το πετύχουμε. Τώρα, όταν έχουμε διασυνοριακά προγράμματα θα πρέπει να ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και τα διάφορα μέσα ε, χρηματοδότησης τα λαμβάνουν αυτά υπόψη, αλλά υπάρχει και πολιτική πίεση ε, σε όλους τους υπουργούς μεταφορών που δεν βλάπτει να τους πιέσουμε, ιδιαίτερα μια που έχουμε διάφορα έργα υποδομών και επέκτασής τους στα κράτη-μέλη να ακουστεί και η δική μας φωνή. Βέβαια, τα προβλήματα αυτά τα διασυνοριακά, ακόμα και αν δεν αρέσει τα κράτη-μέλη, είναι μεγάλα και δεν είναι χτεσινά εδώ και καιρό. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά λοιπόν πολύ εντατικά. Ε, υπάρχουν και προβλήματα με τη μόχλευση τι θα γίνει, ε, θα μετράμε ε, στατιστικές, επιβάτες, μεταφορές. Ε, πάση περιπτώσει, ε, με τροπολογίες σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες έφεραν και το θέμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών, των drones. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα, πρέπει, και θα μπορέσουμε πιστεύω να βρούμε ένα συμβιβασμό πέρα από κόμματα και πολιτικές ομάδες. Το είπα και την τελευταία φορά, το θέμα αυτό με τις εξαιρέσεις από το ε, σύμφωνο σταθερότητα, τα κριτήρια για τις επενδυτικές. Ε, δεν συμφωνώ. Όταν αυξάνει το χρέος δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι καλύτερες οι υποδομές. Θα πρέπει να βρεθεί κάποια συνένεση ή μπορεί και όχι. Χάρηκα πάρα πολύ σε αντίθεση με άλλες εκθέσεις επικεντρωνόμαστε στο θέμα, στην κεντρική ουσία και δεν προσπαθούμε να κάνουμε μικροπολιτική. Ευχαριστώ. Η Σάσκουν Μπιλμπάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Έχει και πάρα πολλή δουλειά. 210 τροπολογίες να επεξεργαστεί. Προσπαθεί να πετύχει συμφωνίες. Πραγματικά έχει πάρα πολλή δουλειά και την ευχαριστώ γι' αυτό. Εγώ θα επικεντρωθώ στις 14 βασικά τροπολογίες που καταθέσαμε εμείς οι φιλελεύθεροι ε, και ε, έχει τα εξής βασικά. Πρώτον, θα πρέπει στον τομέα αυτό να προχωρήσουμε στη ψηφιακή εποχή και σε αυτό τον τομέα, να ενισχύσουμε τη χρήση των νέων τεχνολογιών με την εφαρμογή της καινοτομίας, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι βασικό στοιχείο θεμελιώδες έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των εργαζομένων στις μεταφορές, να βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των μεταφορών και επίσης να προχωρήσουμε στη μείωση ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και είναι και όφελος αυτό για το περιβάλλον. Δεύτερον, οι τροπολογίες ζητούν συνοχή. Ε, το 2013 κάναμε μια αναθεώρηση των ε, περιοτήτων και των ε, ευρωπαϊκών ε, προγραμμάτων. Τρία χρόνια αργότερα δεν είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι γιατί κάθε κράτος μέλος κάνει ό,τι του καπνίσει και δεν έχουμε καμία δυνατότητα ε, που να υποχρεώνει τα κράτη-μέλη μετά από την αναθεώρηση του 2013. Δεν είναι δεσμευτικά. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και τίποτα κυρώσεις έτσι ώστε να εκτελούν τα προγράμματα που είναι από το 1994 υποτίθεται προτεραιότητα ε, κάποια έργα τα οποία τα κράτη-μέλη δεν τα υλοποιούν. Δύο κεντρικές ιδέες λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή και εμείς θα ήμασταν δύο τεθειμένοι να συμφωνήσουμε. Ε, όπως ζήτησε η ε, να υπάρχει μια συνοχή των εθνικών προγραμμάτων με τα ευρωπαϊκά. Γιατί σήμερα το πρωί το είδαμε ξανά. Η επανάπτυξη του τρένου ε, Πού οδηγεί. Στον τουρισμό και στις μεταφορές τα περισσότερα γίνονται από το, ε, και με το αεροπλάνο. Και τι κάνει το αεροπλάνο, ρηπαίνει περισσότερο. Θα πρέπει να απαιτήσουμε ε, συνοχή και συνέπεια στη διάθεση της εισηγήτριας για να προχωρήσουμε, να συμφωνήσουμε και η έκθεσή μας να είναι συνενετική, να είναι πρακτική και αποτελεσματική κυρίως όμως. Ευχαριστώ πολύ. εγώ ευχαριστώ η Μαρία Κύλωνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή, την εισηγήτρια, για το πολύ καλό σχέδιο. Έχω αποβάλει κάμπους αστροπολογίες. Η βασικότερη αφορά τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ε, κατάσταση που διαμορφώνεται μετά τη Συμφωνία των Παρισιών. βλέπουμε τη χρήση των κονδυλίων ε, με έναν τρόπο τελείω διαφορετικό. Η απαλλαγή από τον άνθρακα και σχετική στόχη θα πρέπει να είναι η πρώτη μα προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να κατευθύνουμε το δημόσιο χρήμα σε έργα που μπορεί να επιταχύνουν τι κλιματικέ αλλαγέ. Και αυτό βεβαίω πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλε τι πολιτικέ TNT. Η κατανομή κονδυλίων στην Ευρώπη πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα βελτιώσει τη ζωή των μελλοντικών γενεών. είναι κάτι που ίσως δεν μπορούν τώρα να αντιληφθούν ε, οι σημερινοί ηθήνοντες. Ε, πρέπει όμως ε, να μην αφαιθούμε σε αυτό το είδος την παρέτηση, αλλά να δείξουμε τόλμη και να μην σκεφτόμαστε μόνο του εαυτού μα, να δώσουμε ελπίδα και στι μελλοντικέ γενιέ. Ευχαριστούμε, κυρία Ντελή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Όταν κοίταξα την έκθεση, αναρωτήθηκα τα εξής. Πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτά τα βιώσιμα logistics. Και τι είναι αυτό το πολυτροπικό, δηλαδή τα διάφορα μέσα ε, τα οποία αναφέρονται. Αυτό το βιώσιμο λοιπόν σε σχέση με το ε, logistics τι είναι, είναι χαμηλών εκπομπών άνθρακα και για ό,τι κάνει συνδυασμένες ε, μεταφορές, δηλαδή φεύγουμε από τις οδικές και πάμε σε λιγότερο ρηπαρές όπως για παράδειγμα οι σιδερόδρομοι. Νομίζω ότι αν ακολουθήσουμε αυτό το συλλογισμό θα φτάσουμε πολύ μακριά. Να σας υπενθυμίσω πως το Σεπτέμβριο εγώ ε, ετοίμασα μία έκθεση στο Στρασβούργο μαζί με την Επιτροπή για το Περιβάλλον μία έκθεση στην οποία βλέπε κανείς δύο φορτηγά, το νέο μοντέλο και το μοντέλο το 20 ετια και η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών μοντέλων φορτηγών είναι η διαφορά που έχουμε στην ενεργειακή απόδοση των δύο φορτηγών που ήταν στα του 3%. Δηλαδή ουσιαστικά καμία πρόοδος για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ενώ σε άλλους κλάδους έχει ήδη ξεκινήσει η τεχνολογική μετάβαση και όταν μιλάμε για Logistics να σας πω πως καμία πρόοδος εκεί δεν έχει επιτευχθεί. Άρα λοιπόν στην έκθεσή μας θα πρέπει να έχουμε κανόνες και για τα φορτηγά και για τις δημόσιες πολιτικές που επενδύουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες και νομίζω πια έφτασε η ώρα η Ευρώπη να έχει ένα πραγματικό ε, καθεστώς για τα logistics των πόλεων τουλάχιστον με καινοτόμες και τις καινοτόμες λύσεις όπως για παράδειγμα το cargo pooling στους δρόμους και να προσπαθήσουμε με τον τρόπο αυτό να μειώσουμε το περιβαλλοντορικό κόστος και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη ε, διασυνδεσιμότητα μεταξύ μεγάλων βιομηχανικών περιοχών ε, και σιδηροδρομικών κόμβων. Και αυτά να τα δούμε με το πνεύμα του συμβιβασμού, γιατί δεν έχουμε, αν δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο οδικό χάρτη για το θέμα αυτό, νομίζω πως τα επόμενα χρόνια δεν θα σημειώσουμε καμία πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, διότι καθυστέρησα. Έπρεπε όμως να λάβω το λόγο και στην Επιτροπή Μεταφορών. Ξέρετε, είναι δύσκολο να τα καταφέρει όλα κανείς. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της, διότι η έκθεση αυτή είναι άκρο σημαντική. Η την εφοδιαστική στον τομέα των μεταφορών τη θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική. Και θα πρέπει να έχουμε εθνικές πολιτικές στα πλαίσια των ε, διευρωπαϊκών δικτύων, αλλά να σεβαστούμε και την αρχή της επικουρικότητας, διότι μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές σε ό,τι αφορά τους προσανατολισμούς μας και τα κοινά μας συμφέροντα. Η έκθεση αυτή αναφέρεται και στο πρόγραμμα Γαλιλαίο, ε, προσπαθώντας να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτού του προγράμματος, του τεράστιου δυναμικού που προσφέρεται και στην ε, συνεισφορά μας προς τις διάφορες λύσεις που προτείνονται πάντοτε με πλήρη σεβασμό του περιβάλλοντος. Οι τροπολογίε που προτάθηκαν ε, ε, έχουν να κάνουν και με το κοινωνικό dumping στον τομέα των μεταφορών, διότι πολλές φορές εδώ ε, συγκαλύπτεται ο προστατευτισμός. Ο προστατευτισμός που αντίκειται στην αρχή της ενιαίας αγορά στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον, την εισηγητρία και είμαι στη διάθεσή της για να συντάξουμε συμβαστικές τροπολογίες που θα επιτρέψουν να οδηγηθούμε σε πέρα στο επίπεδο της Επιτροπής. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη, διότι καταλαβαίνω ότι είχατε δειξοδικότατη παρουσίαση από την Επιτροπή όταν υποβλήθηκε η έκθεση αρχικά, οπότε δεν θα τα επαναλάβω όλα. Απλώς να ξεκινήσω λέγοντας ότι το γεγονός ότι υποβλήθηκαν 200 τροπολογίες δείχνει την ιδιαίτερη προσοχή και που προσελκύει η έκθεση αυτή και το θέμα της εφοδιαστικής ε, και των ε, συνδυασμένων μεταφορών σε αυτήν την Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι θα μας βοηθήσετε το θέμα αυτό να το προβάλλουμε επαρκώς και όταν ε, συζητούμε τους διάφορους τρόπους μεταφορών και τους αλληλοσχετισμούς τους. Διότι είναι ένα θέμα περίπλοκο. έχει πάντοτε ένα σωρό ενδιαφερόμενους και ανθρώπους ε, που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Είναι στο κέντρο της προσοχής του κοινού. Καλωσορίζουμε λοιπόν την έκθεση της κυρίας Αγιάλα Ζέντερ και ως προς τις τροπολογίες θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που είναι τα πλέον σκόπιμα για το θέμα της εφοδιαστικής. Θα γνωρίζετε ότι έχουμε ετοιμάσει ένα issue paper, δύο από τους συντονιστές των δικτύων TNT, για την ε, λεγόμενη πολυτροπικότητα, του συνδυασμού δηλαδή των διαφορετικών τρόπων μεταφορών και την εφοδιαστική. Πολλές από τις τροπολογίες που υποβάλλατε ε, στρέφονται και προς την ανάγκη ψηφιοποίησης, απαλλαγής από τον άνθρακα ε, ως προς την εφοδιαστική και το τι αντίκτυπο μπορεί να έχει εφοδιαστική ακριβώς την πολιτική της απαλλαγής από τον άνθρακα και το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πετύχει τα αποτελέσματα τη Συμφωνία των Παρισιών, τη COP21, αλλά και τι ε, επιχειρηματικέ πτυχέ τη ευρωπαϊκή οικονομία και τη βιομηχανία. Αυτό είναι κάτι που θα σα το επισημάνουν ξανά οι συντονιστέ ε, των TNT και του χρόνου. Εμεί την σημασία τη εφοδιαστικής την έχουμε αναγνωρίσει συμπεριλαμβάνοντά την στις υπηρεσίες εμπορίας, εμπορικών μεταφορών και ελπίζουμε ότι με την δική σας την έκθεση θα μπορέσουμε και τις εμπορικές μεταφορές με συνδυασμό διαφορετικών τρόπων μεταφορών να την προωθήσουμε. Ο καλός συνδυασμός των διαφορών τρόπων μεταφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει. Τώρα για την εισηγήτρια που θα πρέπει να καλύψει τόσες πολλές τροπολογίες τόσο διαφορετικού περιεχομένου. Ε, θέλουμε να πούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πλευρά της ότι ελπίζουμε στις συμβαστικές τροπολογίες να καλύψετε όλες τις προθέσεις όλων των μελών της Επιτροπής σας. Ευχαριστούμε και πάλι κυρία Γιάννα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, όπως επίσης και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για όλα τα στοιχεία που ενισχύουν και βελτιώνουν την πρόταση αυτή. Βεβαίως θα ήθελα να καθησυχάσω και τις συναδέλφους που μίλησαν για το κομμάτι που έχει να κάνει με την τεχνολογική καινοτομία γιατί μέσω της ε, ψηφιοποίησης νομίζω ότι θα μπορέσουμε τουλάχιστον να βελτιώσουμε και να μειώσουμε το γραφειοκρατικό βάρος και το, την περιβαλλοντική επίπτωση που έχουν όλες αυτές οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, των logistics μας δηλαδή και να σας πω πως τα κράτη-μέλη τη στιγμή που σχεδιάζουν και θα εφαρμόσουν όλα αυτά σε εθνικό επίπεδο πολύ συχνά έχουν ανακαλύψει πως υπάρχει μια έλλειψη ε, προσαρμογής γιατί αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί να χρηματοδοτηθούν από το Συμβούλιο πολλές φορές δεν έχουν γίνει με έναν τρόπο που να είναι είτε αποτρεπτικός είτε πιστικός για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο μπορούμε αυτή η νέα βάση που εσείς έχετε δίκιο. Είναι ο συνδυασμός της COP21 ε, και των στόχων εκεί για το πώς μπορούμε να μειώσουμε το κόστος της, των εμπορικών μεταφορών έτσι ώστε να έχουν ελάχιστη επίπτωση στο περιβάλλον. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Έχουμε μια σειρά προτάσεων εδώ και θα καθίσω μαζί σας να δω πώς μπορώ να βελτιώσω την πρόταση με τις ιδέες σας, τις οποίες βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα στις 5 Δεκεμβρίου. Επόμενο θέμα ετήσια έκθεση σχετικά με τι χρηματοδοτικέ δραστηριότητε Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εισηγητή είναι ο κ. Μπόγκουσλαφ Λιμπεράτσκι. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχά, να τονίσω ότι μάλλον δεν θα είναι εμφυλεγόμενη η έκθεσή μου. Και δεν θα μα πάρει πολύ χρόνο. Σα παρακαλώ, ησυχάστε. Διότι αλλιώ δεν μπορεί να μιλήσει ο Μιλάμε για χρήμα μία και μόνη τράπεζα. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγο εδώ να υπάρξουν αντιπαραθέσει. Ένα τακί. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε περίπου 80 τροπολογίε, τι οποίε έχουμε εξετάσει με τους και όδη. Του ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία του, όλου και όλε. Έχουμε ετοιμάσει 7 συμβαστικέ, οι οποίε καλύπτουν 50 επιμέρου τροπολογίε. οπότε εν τέλει δεν θα έχουμε τόσε πολλέ τροπολογίε να ψηφίσουμε ιδιαίτερος να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον κύριο Ρικέ, την κύριο Τζίλερ, την κυρία Τελίτσκα, τον, την κυρία Ντελή και πιστεύω ότι έχετε τα έγγραφα μπροστά σας. Δεν θα πω περισσότερα στην πρώτη μου παρέμβαση. Εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια, ευχαρίστως να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ και τη γραμματεία. Ο Ραντεκ να κάνει πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, uh, uh, uh, Θα ήθελα να ξεκινήσω και εγώ με ευχαριστίες προς τον εισηγητή. Τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια και τις τοπολογίες που εγώ υπέβαλα και την καλή σας δουλειά για την ε, έκθεση αυτή, την γνωμοδότηση. Η έκθεση είναι αρκετά ισόρροπη Και το πρώτο θέμα είναι η έκθεση της ΕΤΕ και στοιχεία που έχω θίξει στις τροπολογίες μου. Τα συζητήσαμε μόλις τώρα και με τον κύριο Κατάινεν. Θα συνεχίσουμε με την σχετική γνωμοδότηση για το ΕΦΣΙ να κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λιμπεράτση και για όλη σας τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, Θα είμαι και εγώ το ίδιο συνοπτικός όσο και εισηγητής και ο συναδελφός μου Ρόμπερτ. Να ευχαριστήσω τον Μπόγκοσλαβ για την τόσο καλή του έκθεση, για τη συνεργασία μας. Δεν συμφωνώ. Όταν λέει ότι όταν μιλάμε για χρήμα δεν υπάρχουν διαφωνίες, ίσα ίσα. Το χρήμα προκαλεί πολλούς τριγμούς και συζητήσεις. Όμως εδώ συμφωνούμε σε πολλά. Οι επιπλέον συζητήσεις που είχαμε πραγματικά μας ε, διαφώτισαν περαιτέρω, οπότε νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι όλοι με το αποτέλεσμα της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η Μερία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, πολύ καλή δουλειά του. Λίγα μόνο σχόλια. Και εγώ υπέβαλα τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί επαναλαμβάνω σαν αυτόματο την Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα και τα μέτρα που πρέπει να προβλέψουμε ως αποτέλεσμα αυτής στο μέλλον θα πρέπει να είναι στοχευμένα τα μέτρα που προβλέπουμε, να θέτουν συγκεκριμένου στόχου δηλαδή. Και όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕ, ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι πραγματικά ήλπιζα σύντομα να άλλαζε η συλλογιστική και η προσέγγιση μα. Να μην μιλάμε για τι υποδομέ των μεταφορών σαν ανημονή λύση. Ήλπιζα να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε με τι υπάρχουσε υποδομέ και να αναπτύξουμε, να κάνουμε πιο αποδοτικό τον τρόπο που λειτουργεί το δίκτυο των μεταφορών. Αυτοματοποίηση, κάτι που γρήγορα προχωράει, ψηφιοποίηση. Η δική μου η θεωρία είναι ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε περιτά ε, περιτές ή άστοχες επενδύσεις, γιατί βασιζόμαστε σε υποθέσεις τη τωρινή περίοδου για του διαφορού τρόπου μεταφορών. Γι' αυτό λοιπόν επέμενα στο σχέδιο έκθεση να μην μιλάμε μόνο για τι υποδομέ μεταφορών, αλλά και για τι υπηρεσίε μεταφορών ε, που την ευρύτερη έννοια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η Μαντελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα μου χρειάζεται την ικανοποίησή τη για την ομάδα αυτή και να συγχαρώ τον ε, εισηγητή και να τον ευχαριστήσω για την τόσο καλή μα συνεργασία. Να πω ότι η έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνει πολύ καλέ συμβαστικέ λύσει και εν τέλει πραγματικά δίνει ένα πραγματικό ε, χάρτη, ένα πραγματικό φύλλο για την στην ΕΤΕ. Το είπαμε προηγουμένω και στον κύριο Κατάιναν. Η έκθεση αυτή επαναλαμβάνει προ την ΕΤΕ ποιε είναι οι σωστέ προτεραιότητε. Βλέπουμε την ε, βιώσιμη κινητικότητα, το κλίμα, την ασφάλεια και την κοινοτομία να θέλουμε να την προωθήσουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγο να έχουμε αντίρρηση στην έκθεση αυτό. γύρω και πάλι τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Μπαχ, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστούμε, Μπόγουσλαβ. Ε, διαπιστώσαμε ότι εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά και εντατικά για το θέμα αυτό οι συμβαστικές προτάσεις 7 των αριθμών μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Παρόλο που έχουν γίνει γενναίες επενδύσεις εδώ και δεκαετίες στις μεταφορές, απομένει ακόμα πάρα πολλή δουλειά. Και η έκθεση αυτή πραγματικά αναδεικνύει τα σημαντικότερα σημεία, καινοτόμες διατρο... συνδεδεμένες μεταφορές, ε, γεωγραφική ε, κατανομή, ε, στόχοι ε, της COP21, της Συμφωνίας για το Κλίμα, όλα αυτά τα τονίζει πάρα πολύ ωραία ο, ο εισηγητής. Και η έκθεση συμπληρώθηκε και εμπλουτίστηκε από τους διαφόρους βουλευτές με τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε και πάλι τον εισηγητή για τη συνεργασία. Ευχαριστώ, η κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρεμβαίνω και εγώ για να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης Πρόκειται για κονδύλια και επενδύσει και θα μπορούσαν να υπάρχουν αντιπαραθέσει. Εδώ όμω καταλήξαμε πραγματικά σε μια κοινή γραμμή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι το όντι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, σε μια θετική πορεία. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή που έλαβε υπόψη κάποιε από τι προτάσει μα, όλο ιδιαίτερε αυτέ που έχουν να κάνουν με το ε, δίκτυο των TNT, των Ευρωπαϊκών Δικτύων συνολικά, που είναι πολύ σημαντικά για τη διασύνδεση τη Ευρώπη, αναγνωρίζοντα βεβαίω ότι ακόμη πρέπει να γίνουν επιπλέον προσπάθειε. Ευχαριστώ επίσης που έλαβε υπόψη όλους τους τρόπους μεταφορών όταν Μιλάμε για τα ελαστικά στην περίπτωση των πηγών ρήπανση, αλλά και των διαφόρων διευκολύσεων που όπως ξέρουμε έχουν κάπως ε, αλλάξει κατεύθυνση. Εδώ λοιπόν θέλουμε να φροντίσουμε το που κατευθύνονται οι επενδύσεις καλύτερα ώστε και το ΕΦΣΥ να επιτρέψει να γίνουν επενδύσεις σε αυτό το τομέα ιδίως όταν αφορά τις δημόσιες μεταφορές. Επίσης, για το σύστημα μεταφορών για τους επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μαντέο Ρίτσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους σας της Επιτροπή. Δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Συντομότατος. Ευχαριστώ. Και τώρα ξανά ο Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Υπόθηκαν τα πάντα. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και πραγματικά ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και την ψηφοφορία. Ευχαριστώ τους πάντες, με αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκα, τους Κιώδης δηλαδή κυρίως. Και πραγματικά με ικανοποιεί ιδιαίτερα αυτό που αναφέρατε, ότι αυτά που θέλατε έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση. Χαίρομαι πολύ που εκτιμήσατε την ε, δουλειά μας. Ο καθένας και κάθε μια από εσάς ξεχωριστά. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την τόσο σύντομη παρέμβασή της που ε, περασπίζεται την θέση τη και ευχαριστώ και εσά Πρόεδρε, σα ευχαριστώ όλου. Ευχαριστώ πολύ ψηφοφορία, θα γίνει αύριο. Προχωρούμε. Σημείο 12. Κανόνες αστικού δικαίου σχετικά με τη ρομποτική. Είναι γνωμοδότηση δική μας προς την ε, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, Γεωργ Μάιερ ο εισηγητής, τον οποίο εκπροσωπεί όμως η κυρία Γιούτο. Όχι, Αρνοτσού. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω καταρχήν ε, να σας ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Μάγερ γιατί δυστυχώς δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα να σας πω ως εισαγωγή πως λυπάμαι πολύ λίγο πως ε, μια χούφτα ε, ευρωβουλευτές έβαλαν τα συμφέροντα του κλάδους πάνω από αυτά των Ευρωπαίων και αυτή η γνωμοδότηση τελικά έχει απεισχναστεί από οποιαδήποτε ισχύ και Χαίρομαι που τουλάχιστον ήταν λίγοι γιατί οι περισσότεροι δέχονται τους κανόνες της δημοκρατίας και την ε, ε, βούληση των ε, εκλογέων τους και ξέρουν πως αυτά τα κομματικά τερτύπια δεν ικανοποιούν κανέναν. Λοιπόν, να σας πω πως ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις σας στις τροπολογίες συμβιβαστικές που έχουν λάβει υπόψη ε, αυτά που μας ζήτησε η ECR, η ALDE και το ELK και έτσι έχουμε καταλήξει σε ένα κείμενο ισορροπημένο. Έχουμε ένα συνεπή ορισμό όλων των μέσων συγκοινωνίας ή μεταφοράς με έναν τρόπο σωστό και δυστυχώς αυτό που δεν μπορέσαμε να βάλουμε στο συμβιβασμό είναι ένα κείμενο το οποίο θα ήθελε ο κύριος Μάγερ να έχει καταφέρει να ε, συμπεριλάβει έτσι ώστε χωρίς κομματικούς χρωματισμούς να υπερψηφίσουμε και είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε άλλο σχόλιο και βεβαίως θα του μεταφέρω όλα τα δικά σας σχόλια πριν ψηφίσουμε αύριο. Ευχαριστώ, ο Λουίς Δεγκράντες Πασκουά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Αρνοτού αντικαθιστά σήμερα τον κύριο Μάιερ, τον εισηγητή. Στην Ισπανία έχουμε μια έκφραση που μπορεί να έχει σημασία, που λέει «Η «Ε, ευγένεια υποχρεώνει». Και απαντώ στα παράπονα και στις καταγγελίες. Έχουμε τεράστιες διαφορές και πάρα πολύ γνωστές με την ομάδα του εισηγητού. Αλλά πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήταν αξιέπαινη η προθυμία του να ακούσει ε, τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Έτσι έχουν τα πράγματα. Για διάφορους λόγους δεν θέλουμε να συμμετέχουμε στο συμβιβασμό, αλλά για να διευκολυνθεί ο συμβιβασμό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το συμπεριψηφίσουμε, γιατί ουσιαστικά είναι αρκετά λογική. Η δική μας θέση έχει ως εξής. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν και διαφυλάσσονται στο συμβασμό προστασία δεδομένων, πνευματική ιδιοκτησία, ε, γενικότερα ζητήματα πληροφορικής. Ε, Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στους ε, ε, κώδικες καινοτομία, ασφάλεια των αυτοκινήτων με αυτόματη οδήγηση χωρίς οδηγό και ευθύνη αστική ε, των νέων εργαλείων ε, και που είναι τόσο αποτελεσματικά αλλά με μεγάλη καινοτομία. Συμπέρασμα. Αν περάσουν οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί μαζί με τους λογικούς συμβιβασμούς, ακόμα και αν δεν συμμετείχαμε στην εκπόνησή τους, θα υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, εκ μέρου του κ. Στανχόπης, ο οποίο ήταν ο Ισκιώδης και ο οποίο έφυγε, όχι για την Ινδία αυτό, αλλά για την Τσεχία, και ο οποίο μου ζήτησε να πω τα όσα είπε και ο κ. Δεγκράντες, ε, η ECR θα στηρίξει αυτού του συμβιβασμού, και μετά Βεβαίω θα στηρίξουμε και τη γνωμοδότηση όταν περάσει από την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Η Μερία Κύλωνε. Με ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή και εγώ για το σχέδιο του κειμένου. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να αποφανθεί για αυτά τα θέματα που είναι πάρα πολύ επίκαιρα κατά τα άλλα. Θα πρέπει να ξέρουμε τι φρονεί η μας Επιτροπή. Το κείμενο είναι καλή βάση, αλλά λείπει ο αντίλογος που θέλουμε εμείς να βάλουμε τις δικές μας τροπολογίες. Θέλω να επικεντρωθώ και σε άλλες ε, ε, πτυχές. Λέει ο Πρόεδρος ότι δεν υπάρχει ε, γαλλική διερμηνία, μάλλον ότι άκουγε ο ίδιος γαλλικά αντί για γερμανικά. Να ξαναρχίσω από την αρχή, λέει κυρία Κίλωνεν. Μάλιστα. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή ε, για την πρότασή του. Είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβουλίο να έχει άποψη για αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ επίκαιρα και πάρα πολύ φλέγοντα. Και θα πρέπει να ξέρουμε τι λέει και η δική μας Επιτροπή Μεταφορών. Το κείμενο είναι μια καλή βάση, αλλά λείπει ε, ε, κάποιο στοιχείο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μιλάμε για αυτόματα αυτοκίνητα ή οχήματα χωρίς οδηγό, γιατί η ρομποτική ε, έχει παρουσία και αλλού ε, στις μεταφορές. Παράδειγμα, υπάρχει αυτόματος πιλότος στα αεροσκάφη ε, ή ε, στα πλοία. Η ρομποτική δεν είναι μόνο ένα αυτοκίνητο που προχωρεί στον δρόμο χωρίς οδηγό. Επιπλέον, η ρομποτική θα μπορούσε να αλλάξει τελείως ε, τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιεί το κλάδο των μεταφορών, με μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον. Μας έχει δείξει η ιστορία ότι οι καινοτομίες είναι πολλές φορές πηγή εμπιστοσύνης, αλλά όχι από την αρχή. Δεν θα πρέπει όμως να έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στην καινοτομία, γιατί και ορισμένες εφευρέσεις δεν βελτίωσαν ακριβώς την κατάσταση ούτε τη ζωή μας. Πάντα θα πρέπει να κοιτάμε διάφορες ε, λύσεις και συνδυασμούς για να προχωρήσουν οι μεταφορές. Για μένα καμιά φορά με ανησυχεί αυτή η εστίαση στην αυτοματοποίηση, ότι είναι μια πανάκια ας πούμε, ότι θα μας λύσει όλα τα προβλήματα της αηφορίας και της βιωσιμότητας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε ένα ευρύ φάσμα επιλογών στη διάθεσή μας και πιθανών λύσεων για να μπορούμε να τις συνδυάζουμε και να προχωρούμε. Θα ήθελα επίσης να πω ότι συζητούμε και τη σημασία εδώ της διεθνούς συνεργασίας Στις Ηνωμένε Πολιτείες έχουν ε, μια στρατηγική για τη ρομποτική, την έχουν δημοσιεύσει και θέλουν τα προβλήματα των μεταφορών, ειδικά των οδικών, να λυθούν με την αυτοματοποίηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, για να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ασία και να κανονίσουμε και τη δική μας πορεία. Αυτό θα έχει σημασία για τη διάδοση, για τη διεύρυνση του ρομπότ και σε σχέση με τα σημερινά μας προβλήματα. Ταυτόχρονα θέλω να επιμείνω στο εξής. Έχουν γίνει μεγάλες τεχνολογικές πρόοδοι και πρέπει να προβλέψουμε τι μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια και μάλιστα τα επόμενα 50 χρόνια. Χρειαζόμαστε νέα προγράμματα μεν, νέα σχέδια, αλλά να ξέρουμε προ ποια κατεύθυνση θέλουμε να πηγαίνουμε. Η δική μα πολιτική ομάδα Γκουε υποστηρίζει την έκθεση αυτή και θα την υπερψηφίσει. Ευχαριστώ, η Καρή Μαντελή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για τη δική μου ομάδα η έκθεση αυτή δημιουργεί προβλήματα γιατί δεν τονίζει επαρκώς το πραγματικό διακύβευμα. Δηλαδή, θα πρέπει να ρωτηθούμε, και είναι καινούργιο το θέμα αυτό, ποια είναι η αστική ευθύνη όταν χρησιμοποιεί κανείς ρομπότ. Η αστική ευθύνη. Και η συνάδελφος, ε, κυρία Κίλονεν, μας είπε πως έχουμε την τάση να μιλάμε μόνο για τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Όχι. Όλα έχουν πολλαπλασιαστεί σίγουρα. Έχουμε και βέβαια τα οχήματα χωρίς οδηγό, αλλά έχουμε και τα drone, τα οποία δημιουργούν πάρα πολλά θέματα. Και όλα τα τηλεκατευθυνόμενα εξ αποστάσεως, που ενδεχομένως μπορεί μετά να παρουσιάσουν και ευφυή συμπεριφορά. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε τι θα γίνει σε περίπτωση ατυχήματος. Είναι απαραίτητο να υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και το οποίο θα ορίζει ποιος φέρει την ευθύνη, ο χρήστης, ο κατασκευαστής, ο χειριστής των δεδομένων, το ίδιο το όχημα, ποιος φέρει μερικά ή ολικά την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτό είναι πραγματικά σπαζοκεφαλιά. Και η απάντηση ακόμα δεν έχει δοθεί. Ούτε στην έκθεση, ούτε κατά τη στιγμή των συζητήσεων, παρόλο που η τεχνολογική εξέλιξη τρέχει. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν και θα πρέπει να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μήνυμα, ένα μήνυμα ισχυρό έτσι ώστε να συζητήσουμε το συντομότερο δυνατόν το θέμα αυτό και να προτείνουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο με μια πρόταση νομοθεσίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε εμείς, γιατί όπως σας είπα η τεχνολογική επανάσταση δεν θα μας περιμένει, θα προχωρήσει πολύ γρήγορα και εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ασφάλεια, ότι υπάρχει ευθύνη για όλα αυτά. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εμείς να προλάβουμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σφαν Μίλτενμπεργκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ε, αρχίσατε νωρίτερα τη συζήτηση από ό,τι προβλέπετε. Η έκθεση αυτή δεν είναι έκθεση, είναι γνωμοδότηση, πλην σημαντικότατη. Ε, ευχαριστώ ε, λοιπόν και είναι σημαντικό να το κοιτάξουμε λίγο, να σταθούμε μια στιγμή. Ε, αυτόματα αυτοκίνητα, καμιά φορά και πλοία, ε, drones, είναι ένα θέμα του μέλλοντος. Και θα περίμενε κανείς να γίνει μια πολύ καλή ανάλυση, οξία ανάλυση, με πάρα πολύ στοχευμένη γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, Γιούρι. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με το συμβιβασμό που έχουμε εδώ ο εισηγητής έβαλε σε ένα μεγάλο τσουβάλι όλες τις τροπολογίες, οι οποίες ήταν πολύ καλές ορισμένες, με πολύ προστιθέμενη ασία και έχει βγάλει ένα συμβιβασμό από 19 τροπολογίες σε ένα σχετικά μικρό συμβιβασμό. Αποτέλεσμα, έχει χαθεί αυτή η οξύτητα, αυτή η ε, κριτική ματιά και υπάρχουν και μεγάλα λάθη, υπάρχουν μεγάλες ε, ανακρίβειες και είναι κρίμα για μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών. Γι' αυτό το λόγο θα ε, πρότεινα και θα προτιμούσα να ψηφίσουμε ξεχωριστά τις τροπολογίες και όχι το συμβιβασμό. Μας έχει ε, απογοητεύσει λίγο η διαδικασία τέλος που δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε με άλλες πολιτικές ομάδες για εναλλακτικέ συμβαστικές τροπολογίες. Σταματώ εδώ. Θα δούμε στην ψηφοφορία τι θα βγει και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Αλεσάνδρος Παρτιρώνη. Okay. Thank uh, uh, say... Θα πω μόνο Δύο λόγια για την έκθεση αυτή. Οι τροπολογίες τούτες. Και θα είμαι σύντομος. Οι τροπολογίες λοιπόν αυτές ή μάλλον να τα αντιστρέψω. Εμείς είμαστε όλοι... Έχουμε αναγνωρίσει όλη τη σημασία των ζητημάτων αυτών, των συμβαστικών τροπολογιών και θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα δούμε στα πλαίσια της ε, σχετικής πλατφόρμας, να δούμε την αστική ευθύνη, να δούμε τι κάνει η DigiGrow, τι σημαίνει ιδιωτικότητα και πρόσβαση σε δεδομένα και μία σειρά θεμάτων που άπτονται αυτών τώρα για την ευθύνη και για την ασφάλεια. Ήμουνα πριν από δύο μέρες, ήμουνα σε μια συνάντηση της Gear 2030 και είδαμε πώς θα επηρεάσουν όλες αυτές οι εξελίξεις στον κλάδο τον ασφαλιστικό. Και επίσης θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτή η οδήγηση χωρίς οδηγό, για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι κομμάτι της βιώσιμης κινητικότητας, που είναι η σφαιρικότερη στρατηγική που επιδιώκουμε στον κλάδο των μεταφορών. Δεδομένου το ότι όταν λέμε αυτόνομο μιλάμε για κάτι το οποίο έχει ράγες, ε, θα μειωθεί η, θα μειωθεί το επίπεδο συμφόρηση, άρα λοιπόν θα έχουμε καλύτερα επίπεδα βιώσιμη κινητικότητας. Και έχει γίνει πολλή προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό με αποτελέσματα τα οποία θα δημοσιεύσουμε τις επόμενες εβδομάδες, όπου θα παρουσιαστεί μία ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα, για τα συστήματα συγκοινωνιών ε, στην Ευρώπη, όπου θα έχουμε μία ε, συνεργατικότητα με τις αυτοματοποιημένες μεταφορές και στα πλαίσια της διαδικασίας για το 2030, στα τέλη του 2016 θα παρουσιάσουμε τα πρώτα αποτελέσματα για τα πρώιμα συστήματα, τα συστήματα του 2020 όπως αναφέρονται και θα έχουμε και την ανακοίνωση τη σχετική ε, από το Gear 2030 στις αρχές του 2017, ίσως και λίγο αργότερα. Το 2017 θα κάνουμε και μια διάσκεψη για την συνδεδεμένη και για την αυτοματοποιημένη οδήγηση, έτσι ώστε όλα αυτά να συνδυαστούν μέσα στους ευρύτερους στόχους της μεταφορές και να πω πως και στη Γιούνισε είμαστε δραστήριοι, έτσι ώστε να μην είμαστε μόνο Ευρωπαίοι στα όσα προσπαθούμε, αλλά να ενταχθούμε και στο παγκόσμιο πλαίσιο. Για τον Γαλιλαίο νομίζω πως ε, την σχετική στρατηγική την ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες περίπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ξανά η κυρία Αγνοτού, δεν ξέρω αν θέλει το λόγο. Να. Ακούστε, Πρόεδρε. Σημείωσα όλα τα σχόλια. Ευχαριστώ τους δύο πρώτους ομιλητές και την κυρία Κίλονεν που παρά τις επιφυλάξεις της εκφράστηκε θετικά. κυρία Ντελή, κατάλαβα καλά. Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα της ευθύνη. και ο πρόσωπος Ευρωπαϊκή Επιτροπής δεν το διευκρίνησε, αλλά νομίζω ότι τίθεται επί τα άπητος και προφανώς θα πρέπει να μιλήσουμε για την αστική ευθύνη. Πλην όμως δεν δηλαδή, είναι το παρόντος αυτό και όσο για σας κύριε που συγγνώμη δεν ξέρω και πώς σας λένε, Φαν Μίλτενμπεργκ. Μάλιστα. θα σημειώσω αυτά που λέτε και θα τα διαβάσω στον κύριο Μάιερ. Αλλά εγώ είχα την αίσθηση αντιθέτως ότι στους συμβιβασμούς ε, του κυρίου Μάιερ ε, προσπάθησε και κατέβαλε προσπάθεια δηλαδή ουσιαστική έτσι ώστε βέβαια όσο αυτό ήταν εφικτό, να συγκεράσει τις περισσότερες ιδέες, γιατί έχει πολλέ τροπολογίε. Θα του τα διαβιβάσω, εν πάση περιπτώσει, εξ ονόματό σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και πάμε στο επόμενο θέμα στη μέρη σε διάταξη. Έκθεση εφαρμογή σχετικά με την ίση μεταχείριση στην πρόσβαση αγαθά και υπηρεσίε και την παροχή αυτών. Γνωμοδότηση είναι για έκθεση πρωτοβουλία Επιτροπή Γυναικών. Δικό μου συντάκτη γνωμοδότηση είναι ο Γιάννη Νίλσον, ο οποίο και έχει αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομο. Ξεκινώντα, να πω ότι ε, πολύ καλώ ετοιμάζει αυτή τη γνωμοδότηση η Επιτροπή μα προ την Επιτροπή ε, ΘΑΜ όπως βλέπω, ε, πολλές άλλες επιτροπές ε, απήχαν από το να συντάξουν ομοδότηση. Δεν είναι πολύ καλό αυτό. Η καθήλυνα αρμόδια είναι η Επιτροπή θάμα, αλλά το θέμα είναι πραγματικά οριζόντιο. Δεν μπορεί να μην άπτεται και το τομέα των ανατηφορών για τον οποίο είμαστε εμεί υπεύθυνοι και οι υπόλοιπε επιτροπέ Γιούρι και οι υπόλοιποι νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχουν γνωμοδοτήσει. Η ΙΜΚΟ λόγου χάρη, η ΙΤΡΕ δεν θα έπρεπε να τοποθετηθούν για τα θέματα ισότητα των φύλων. Νομίζω ότι πρόεδρε σωστά το θέσατε όταν ε, συναντηθήκαμε και ε, ήταν πραγματικά πολύ εύστοχη ερώτηση. Τέλο πάντων, να περάσω στην γνωμοδότηση αυτή καθεαυτή. αυτή είναι καλή πρόταση. Υπάρχουν πολλέ τοπολογίε. Είχαμε μια συνάντηση των σχεδόν τώρα και καταλήξαμε σε ένα κείμενο επί το οποίο νομίζω μπορούν να συμφωνήσουν όλοι οι σκιώδει. Ε, είναι πολύ ε, ικανοποιητικό. Μπορώ να συμφωνήσω με τους ε, και τους ευχαριστώ για την συνεργασία του. Το κείμενο είναι ακόμα καλύτερο ε, και μπορούμε να ελπίζουμε σε ευρεία στήριξη για την έκθεση αύριο στις προφορίες. Ευχαριστώ, Ζόρτζου Μπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Νίλσον για την καλή του εργασία και την καλή συνεργασία μαζί μας, τους κοιόδης συγητές. Πολύ αξία, σημείο αξιοσημείωτη. Τα σημαντικότερα σημεία τα έχουμε συμφωνήσει. Να πω κάτι για τον τουρισμό και χαίρομαι που πήγε αυτό και για κάποιες βελτιώσεις στα υγειονομική κατάσταση των εγκαταστάσεων και επίσης ε, αρρωγή και βοήθεια ε, σε περίπτωση επιθέσεων ε, κλοπών, ληστιών κτλ. Ελπίζω αύριο να ψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ, ο Ρόμπερτ Ζήλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω σχόλια. Καλώ Η Γκεζίνα ναι. Κρίμα, Ρόμπερτ. Γιατί αφορά και άνδρες αυτό το θέμα. Ε, το να ε, είναι εντάξει οι γυναίκε και να έχουν την ίδια πρόσβαση. Ναι, πραγματικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εφαρμοστεί μια οδηγία έτσι ώστε οι γυναίκες να έχουν ίση πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, να το ελέγχει ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα η Επιτροπή Γυναικών ε, έχει επιληφθεί ε, του θέματος ε, αυτού και θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν και άλλες επιτροπές. Δεν είναι πάρα πολύ για μας αυτό το θέμα, αλλά ας πούμε να μην είναι πιο ακριβή η ασφάλεια σε περίπτωση ταξιδίων για τις έγκυες γυναίκες. Αν λέμε ότι δεν κάνουμε παιδιά, θα τις επιβαρύνουμε και οικονομικά με έγκυες και θέλουν να ταξιδέψουν. Είχαμε μεγάλη συμφωνία, μεγάλη στην αντίληψη. Ελπίζω αύριο να περάσουν όλες οι συμβαστικές τροπολογίες. Μπορεί να διαφέρουμε σε μερικές λεπτομέρειες, αλλά σε γενικές γραμμές είναι καλή γνωμοδότηση. Και χαίρομαι που η Επιτροπή Μεταφορών δεν απέφυγε να γνωμοδοτήσει για ένα τέτοιο θέμα. Ευχαριστώ η κυρία Κίλωνεν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πρόταση αυτή και ευχαριστώ πολύ και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Θα πρέπει να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και εγώ πρέπει να σου πω πως χάρηκα ιδιαίτερα που η Επιτροπή Μεταφορών συνέταξε μία γνωμοδότηση γιατί για τη δική μου ομάδα ήταν σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε ε, για τη βία κατά των γυναικών που θα θέλαμε να εξαλειφθεί από τα μέσα μεταφοράς και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και το θέμα της απασχολησιμότητας των γυναικών που θα πρέπει να βελτιωθεί ε, στο χώρο των ε, μεταφορών και να σας πω επίσης πως δεν πρόκειται με τον τρόπο αυτό να αυξήσουμε ε, την ισότητα αν δεν αναλάβουμε και δράση. Γιατί μόνο με γνωμοδοτήσεις δεν θα τα καταφέρουμε. Δράσεις οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν δράσεις οι οποίες θα βελτιώσουν τις εργασιακές συνθήκες έτσι ώστε να είναι όλα πιο ελκυστικά για τους εργαζόμενους και κυρίως για τις γυναίκες. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον συνάδελφο, ήταν πολύ επικοδομητική προσπάθεια που έκανε και πραγματικά τα πήγαμε καλά και με σένα και με όλους ε, στην ομάδα γιατί δεν εργάζονται βέβαια μόνο οι βουλευτές εδώ, ε, ε, οι βουλευτές μόνο, έχουμε και μια ολόκληρη ομάδα. Κυρία Ντελή παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Πήρα το λόγο ε, εκ μέρους ε, συναδέλφου που δεν παραβρίσκεται σήμερα. Η γνωμοδότηση είναι καλή. Είναι καλό που δίδεται αυτή η μάχη κατά των διακρίσεων που επηρεάζουν τις γυναίκες και καλό θα ήταν να αποδείξουμε πως η θέση της γυναίκες σε επίπεδο ασφάλειας, ε, σε κατά πόσο κινδυνεύει στο χώρο των μεταφορών είναι θέματα που θα έπρεπε να μας απασχολούν και έχουν εμπίσει τροπολογίες. Οπότε εμείς θα υπερψηφίσουμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρή Κριστίνα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά και για την εργασία σας. Αλλά κοιτάξτε να δείτε εγώ, βέβαια δεν σας εκπλήξει, δεν το βλέπω καθόλου με τον ίδιο τρόπο το ύφο τη έκθεση και ακόμα περισσότερο των τροπολογιών που προτείνουν κάποιοι συνάδελφοι με κάνουν να είμαι πάρα πολύ καχύποπτη γιατί σήμερα ο μόνος ανυπέρβλητος ορίζοντας ε, στη ε, θεσμικά όργανα των Βρυξελών είναι να εξαλειφθούν οι ανθρωπολογικέ διαφορέ μεταξύ των δύο φύλων ή να καταπολεμηθεί το περίφημο στερεότυπο των ε, φύλων. Μα άνδρες γυναίκες είναι ίσοι είτε απέναντι στον νόμο είτε απέναντι στους μισθούς που εκεί κι αν είναι πρόβλημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά, γιατί ε, πραγματικά ταλαιπωρείται και στραπατσάρεται. Τώρα το διαβάζετε με ιδεολογικό τρόπο παντού, ε, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορών που βλέπουμε σήμερα, σε τέτοιο βαθμό που θα πρέπει κανείς να απελπίζεται δηλαδή που δεν υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που να οδηγούν μετρό φορτηγά ή ε, να ε, είναι σε χειρονακτικές εργασίες. Άρα ακόμα περισσότερο να μπλέκεται το ευρωπαϊκό επίπεδο στα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ζητήματα, περιφρονώντας ε, κάθε αρχή επικουρικότητας που θυμίζω ήταν και στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Πραγματικά τα διαβάζω πολλές φορές και εκπλήσωμαι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει δεν έχει αρκετά προγράμματα, ε, εντολές και τα λοιπά, ε, θετικές ως προς το, προς το φύλλο. Δηλαδή μεταφορές να είναι ουδέτερες ως προς το φύλλο εντός εισαγωγικών ή χωρίς αποκλεισμούς. Ανεξαρτήτως φύλλου. Μα δεν καταλαβαίνω γρή και διαβάζω μια άλλη τροπολογία που ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να προωθήσουν και να υποστηρίζουν τη χρήση του ποδηλάτου. Του ποδηλάτου. Άκουσαν, άκουσαν και ιδιαίτερα για τις γυναίκες των οποίων ε, η πολιτιστική, η θρησκευτική ε, προέλευση, η ανδροκεντρική νοοτροπία δεν τη σωθεί προς το ποδήλατο. Πραγματικά πρέπει να το διαβάσω περισσότερες φορές για να καταλάβω τι εννοεί εδώ ο ποιητής. Μήπως θέλετε να πείτε ότι είναι σύμβατος ο Ισλαμικός νόμος με τις ευρωπαϊκές αξίες και δεν το λέτε. Και πώς θα λυθεί το πρόβλημα Ισλαμοποίησης των κρατών μας. Τελευταίο. Αυτή η ορολογία καμιά φορά είναι εξωφρενική. Ε, προβλήματα λέτε ανασφάλειας στις συγκοινωνίες, στις δημόσιες. Πολύ ωραία. Αλλά διαβάζοντας μερικά, για να το λύσουμε αυτό, φαίνεται ότι αρχή, αρκεί να δούμε ποιο έχει την ευθύνη. για να υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές, γιατί υπάρχει πρόβλημα, ε, εγκληματικότητας πρέπει να το καταλάβουμε και να παραδεχθούμε ότι οι πολιτικές που υιοθέτησαν ε, οι διαδοχικές κυβερνήσεις και η χαλάρωση της δικαιοσύνης σε πολλά κράτη-μέλη και η αδράνεια ε, είναι που ευθύνονται και δεν θα λυθούν αυτά με τέτοιου είδους ιδεολογικά φορτισμένες εκθέσεις και μιλώ για την έκθεση της Επιτροπής Γυναικών που θα καταφέρουμε να λύσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μάρβιν Λεπούλ από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε Γενική Διεύθυνση Just. Δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Θα μιλήσω εγώ εκ μέρους τους ε, και ζητώ και συγγνώμη εκ μέρους τους. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας που ασχολείται με το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και καλωσορίζουμε το γεγονό ότι ασχολείστε ως προς την υλοποίηση της οδηγίας να διευκρινίσουμε ότι όλα τα μέλη έχουν λάβει μέτρα για την υλοποίηση της οδηγίας και παρομοίως σε αυτή τη φάση ε, θα έπρεπε, πιστεύουμε, να επικεντρωθούμε στο να υλοποιείται σωστά η οδηγία, στο κατά πόσο υπάρχει συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση. Όσο για το έγγραφο εργασίας, Θα μελετήσουμε προσεκτικά τι προτάσει που θα έρθουν στα χέρια μα από το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νίλσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι η ευθυγράμμιση στις μεταφορές σημαίνει ότι ε, Όλα αυτά αφορούν τα ανθρώπινα όντα ανεξαρτήτως φίλου και όχι άντρες και γυναίκες πλέον. Εδώ και 15 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Οι γυναίκες αποφάσισαν Ε, να τονίσουν το γεγονό ότι πρέπει να ακούμε τι απόψει όλων, όλων των πολιτών, είτε είναι άνδρε είτε γυναίκε. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε και αυτό θέλουμε να θυμόμαστε ότι σημαίνει η ευθυγράμμιση τη διάσταση ε, τη όταση των δύο φύλων. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία όλων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να βελτιωθεί η κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Οπότε και ολοκληρώνεται έτσι η σημερινή μα συνεδρίαση και ακολουθεί και κλεισμένον των θυρών η συνεδρίαση των συντονιστών μας.